Uh, good morning, colleagues. Uh, Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Να ξεκινήσουμε με το σημείο 1 της ημερησίας διάταξης, όπου έχουμε κάποιες αλλαγές. Το σημείο 8 για την ε, εξέταση των τροπολογιών για το, το Ταμείο Συντερικής Ασφάλειας θα ήταν ε, η συγκήτριά μας η κυρία Χολμάιρ θα αναβληθεί για τις 24 ε, Ιανουαρίου. Έχουμε ένα νέο σημείο 8. Θα εξετάσουμε τις τροπολογίες για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου αξιωματικών σύνδεσης. Η συγκίτρια είναι η κυρία Κιέγκε. Θα αντικαταστήσει λοιπόν το άλλο 8 για το 25 η ψηφοφορία για το θέμα της προενταξιακής ε, έχει αναβληθεί για τις 23 ε, και το 30 η ψηφοφορία για τις διοργανικές ε, διαπραγματεύσεις για τις ε, πρόδρομες ουσίες για τα κριτικά θα γίνει μετά το 1933. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις σε αυτά, εγκρίνεται η τροποποιηθή σε ημερήσια διάταξη. Έγκριση των πρακτικών τη 31η Αυγούστου και της 15η Ιανουαρίου και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, εγκρίνονται. Και γλώσσε. Έχουμε διερμηνία σε όλε τι γλώσσε εκτό από τα Δανέζικα, τα Κροατικά και τα Γοϊδελικά και έχω διάφορες ε, ανακοινώσεις για τις κατεξοδότηση πράξεις. Θα τα διαβάσω όλα αυτά πάλι. Λοιπόν, συγγνώμη, θα σας βασανίσω με, με τις συνήθεις ε, κατεξοδότηση και εφαρμοστικές πράξεις. Πρέπει να το κάνω από ό,τι φαίνεται. Οπότε, οι κατεξοδότηση και εφαρμοστικές πράξεις εφαρμοστικές στις 9 Ιανουαρίου το Κοινοβούλιο έλαβε το σχέδιο της εφαρμοστικής απόφασης και τα παραρτήματα για την χρήση των προσωπικών στοιχείων και των δακτυλικών αποτυπωμάτων και τα άλλα στοιχεία. Η βασική πράξη είναι ο κανονισμός 2017-2026-30 Νοεμβρίου για τη δημιουργία του συστήματος και την εισαγωγή των στοιχείων για την εγγραφή των στοιχείων για την είσοδο και την έξοδο και την άρνηση εισόδου για την τροποποίηση του συμφωνίας που εφαρμόζει την συμφωνία του Σέγγεν και τους κανονισμούς 767-2008 και 1077-2011. Η, ε, η υποδοχή αυτού του της ε, εφαρμοστική πράξης θα ανακοινωθεί σε όλα τα μέλη της ΛΥΜΠΕ μέσω της, ε, του newsletter στι 11 Ιανουαρίου. Στι 8 Ιανουαρίου το Κοινοβούλιο έλαβε δύο σχέδια εφαρμοστικών αποφάσεων. Το πρώτο έχει να κάνει με τη διατήρηση και την πρόσβαση στο ΕΤΙΑΣ με βάση το κανονισμο 733 b και το κανονισμό 2018-1240 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και δεύτερον για τις τεχνικές λύσεις για τα κεντρικά σημεία πρόσβαση στο κεντρικό σύστημα του ETIAS ε και για μια τεχνική λύση για να διευκολυνθεί η συλλογή των στοιχείων από κράτη-μέλη και το Europol για να δημιουργούνται στατιστικές και την ε, πρόσβαση στο ETIAS ε για εφαρμογή του νόμου με βάση το άρθρο 73.3b του κανονισμού 2018-2240. Το βασική πράξη είναι ο κανονισμός Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τη 12 Σεπτεμβρίου 2018 που δημιουργεί ένα ευρωπαϊκό σύστημα ετιάς και που τροποποιεί τους κανονισμους 1077-2011, 515-2014, 2016-99, 2017 2017-2026 ενημέρωση για αυτές τις εφαρμοστικές πράξεις ε, θα είναι στο newsletter της ΛΥΜΠΕ στις 11 Ιανουαρίου και όποιος έχει θα πρέπει να το κάνει πριν από τις 22 Ιανουαρίου, 12 το μεσημέρι. Και τέλος, 9 Ιανουαρίου το Κοινοβούλιο έλαβε το αναθεωρημένο σχέδιο εφαρμοστικής απόφασης της Κομισιόν για την επαρκή προστασία προσωπικών δεδομένων από την Ιαπωνία, βασική πράξη ο κανονισμος 2016 2016-679 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επαρκή προστασία των προσωπικών δεδομένων από την Ιαπωνία, η ενημέρωση για αυτές τις εφαρμοστικές πράξεις ε, θα ανακοινωθεί στο newsletter της 11 Ιανουαρίου και όποιος έχει αντιρρήσει να το κάνει πριν τις 23 Ιανουαρίου το μεσημέρι. Ωραία. Τώρα, τα θέματά μας σήμερα το πρωί. Καλώς ορίζω τον Σάιμον Μόρντι που είναι ένα πρωτή γενικό διευθυντή τη Γενική Διεύθυνση Home. Ε, Καλώ ήρθε, Σάιμον. Σε ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, στις 10 Δεκεμβρίου η Επιτροπή έδωσε την έγκρισή της στη συμφωνία που ε, συνάψαμε με την Αλβανία. Ήταν η πρώτη συμφωνία αυτού του τύπου, όπως θα θυμάστε. Ο Σάιμον ήταν στην Επιτροπή μας την 1η Φεβρουαρίου πέρυσι για να μας ενημερώσει για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων. Χαιρόμεθα που έχουμε αυτή την ευκαιρία να ακούσουμε για την πρόοδο και τα αποτελέσματα της συνέχισης των διαπραγματεύσεων. Λάβαμε μια, ένα σημείωμα δύο σελίδων από την Επιτροπή. Χαίρομαι πολύ που ο κύριος Σάιμον Μόρντιου είναι εδώ για να μας κάνει μια παρουσίαση. Θα υπάρξει παρουσίαση. Μετά θα μιλήσουν οι σκιώδεις για τις συμφωνίες ε, με την Αλβανία και την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Σάιμον, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και καλή χρονιά σε όλους. Νομίζω ότι η χρονιά αυτή θα είναι αρκετά απαιτητική. Γιατί τα συζητάμε όλα αυτά θα σας πω. Αυτό που διαπιστώσαμε όταν είχαμε την μεταναστευτική κρίση 2015-2016 ήταν ότι οι εταίροι μας και φίλοι στην, στα Δυτικά Βαλκάνια είχαν πολύ μεταναστευτική πίεση και οι η διαδρομή μέσω των Δυτικών Βαλκανίων ήταν ε, η κύρια είσοδο στα Βαλκάνια. Ο Frontex εκείνη την εποχή δεν είχε νομική εντολή για να αναπτύξει σε τρίτη χώρα συνοριοφύλακες. Αυτό ήταν ε, ένα σημαντικό πρόβλημα και έλλειψη. Και γι' αυτό λοιπόν το 2015 προτείναμε να ενισχύσουμε την εντολή της Ευρωπαϊκής Συνοριακής και Ακτοφυλακής, να του δώσουμε δυνατότητα δηλαδή να διεξάγουν κοινέ επιχειρήσεις στην επικράτεια τρίτων χωρών, βεβαίω ε, εφόσον αυτές οι τρεις χώρες συμφωνούν. Αυτή τη δουλειά κάναμε λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο και αρχικά ζητήσαμε από το Συμβούλιο να υπάρξουν διαπραγματεύσει με τη Σερβία και την πήγαμε Δέλτα Μη και κατόπιν σε μια δεύτερη φάση με την Αλβανία, το Μαύρο και την Βοσνία Ζεγοβίνη. Όπως θα γνωρίζετε από τις δικές σας συζητήσεις, οι διαπραγματεύσεις με την πήγα Δελταμή, την Αλβανία πήγαν αρκετά σύντομα. Τα καλά νέα που έχω λοιπόν είναι ότι οι διαπραγματεύσεις για τις ε, συμφωνίες αυτές με όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων ολοκληρώθηκαν επιτυχημένα. Να σας συνοψίσω λοιπόν τις διαπραγματεύσει με τη Σερβία, την, ε, το Μαυροβούνιο και τη Βοσνία Αρζεγοβίνη. Ούτω ή άλλω έχετε μια συνόψηση δύο σελίδων και φυσικά οι συμφωνίες θα σταλούν στην γραμματεία, της, στη γραμματεία σας, όπως κάνουμε συνήθως. Ξεκινάω με τη Σερβία. Οι διαπραγματεύσεις ε, πήραν πολύ χρόνο. Καταλήξαμε σε συμφωνία τέλη Σεπτεμβρίου η οποία συμφωνία έχει ήδη μονογραφηθεί και πριν τα Χριστούγεννα η Επιτροπή ενέκρινε την ε, πρόταση αποφάσεως του Συμβουλίου ούτως ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί με την υπογραφή της αυτή συμφωνία και εφόσον εγκρίνει την απόφαση το Συμβούλιο που αναμένεται τέλη τρέχοντος μηνός η συμφωνία θα υπογραφεί μετά. Από τις προηγούμενες συζητήσεις που είχαν γίνει σας είχα ενημερώσει ότι υπήρξαν δύο δυσχέρειες διαπραγματεύσεις. Πρώτη, κλασική, πώ θα αναφερθούμε στο κοσφοπέλιο. Ε, δεν είναι δυνατόν να έχουμε πολλές φάνταστε λύσεις. Και τελικά έχουμε την ε, στάνταρ ε, υποσημείωση που αναφέρεται στην απόφαση 1244 του 1999 και είχαμε κάποια προβλήματα με τις αποφάσεις ασυλίας η Σερβία δεν ήθελε να δώσει ασυλία τελικά, αλλά τελικά ε, δέχθηκε η Σερβία το συμβασμό που είχαμε με όλε τι άλλε χώρε, την αρχή δηλαδή τη λειτουργική ασυλία. Δηλαδή, εάν ε, συμβεί κάτι κατά της, ε, την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι υπάλληλοι έχουν ασυλία. Και ο εκτελεστικός διευθυντής του οργανισμού αυτού έχει την ευθύνη για να ε, πιστοποιήσει ότι οι πράξεις ε, προέκυψαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων. Και αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν υπόκειται ενδεχομένω στην ε, ποινική δικαιοσύνη της χώρας του. Αυτό είναι μέσα στο περιεχόμενο της συμφωνίας. Με Το Μαυροβούνιο ε, είχαμε περισσότερα προβλήματα και οι φίλοι μα στο Μαυροβούνιο είχαν διάφορα προβλήματα για να το επιβεβαιώσουν πολιτικό επίπεδο. το κείμενο είναι αρκετά ε, σταθερό και ψάχνουμε για ημερομηνία για την μονογραφή. Το κείμενο ε, τη συμφωνία αυτή είναι σαν το πρότυπο για τη γεωγραφικό περιορισμό, τα καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής η μόνη ουσιώδης αλλαγή στη συμφωνία αυτή που ήθελαν ε, αυτοί του Μαυροβουνίου ήταν να τους διαβεβαιώσουμε ότι αν κάτι δεν ε, γίνεται κατά τη διάρκεια των καθηκόντων και ναι μεν ε, και εφόσον βεβαίως οι ομάδες μας, ε, της δικής μας, ε, του δικού μας οργανισμού δεν θεωρείται ότι ενεπλέκοντος αυτήν την ενέργεια θα μπορούσαν να είναι μάρτυρες στα δικαστήρια του Μαυροβουνίου. Με την πήγα Μαδελταμή υπήρχε ένα θέμα, γιατί ήταν πολύ σημαντικό. Γιατί πριν από 20 χρόνια είχε υπάρξει ο τραγικός θάνατος ενός πολίτη τους από ε, έναν στρατιώτη του ΝΑΤΟ, ο οποίος τον χτύπησε με το αυτοκίνητό του και μετά τον βγάλανε γρήγορα από τη χώρα. Και είπαμε ότι θα υπάρχει μία ε, ρήτρα που θα λέει ότι και οι δύο πλευρές δεν θα σπεύσουν να βγάλουν από τη χώρα όποιον έχει ε, ε, υποπέσει σε κάποιο αδίκημα μέχρι να πιστοποιήσει ο υπεύθυνο της υπηρεσίας μας, της υπηρεσίας των, της συνοριοφυλακής, ότι η πράξη αυτή έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων του ή όχι. Με τη Βοσνία Ζεγοβίνη ολοκληρώσαμε τις διαπραγματεύσεις πριν τα Χριστούγεννα και τώρα γίνεται η μονογραφή της. Το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με τη Βοσνία Ζεγοβίνη είναι ότι ήθελαν να επεκταθεί η περιοχή που θα μπορούν να δράσουν αυτές οι ομάδες. Γιατί το καταστατικό της ε, συνοριοφυλακής μας περιορίζει στο να δράσουμε μόνο σε όμορες χώρες με, την, ε, με τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης εκείνη θα ήθελαν να μπορέσει να επεκταθεί και στα σύνορά τους με την Σερβία και την, ε, και την πρώην Ιγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ε, αυτό μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει. Δεν είναι δυνατόν μέχρι στιγμής νομικά. Τι κάναμε λοιπόν, υπογραμμίσαμε ότι θα μπορούσε να υπάρχει μια ρήτρα που να μιλάει για γενική στήριξη μέσω της συνοριοφυλακής με άλλα μέσα πέρα από την ανάπτυξη ομάδων με εκτελεστικές αρμοδιότητες. Κάτι που ήταν ε, λίγο δυσχερές με τους Βόσνιους θέλανε πολύ συγκεκριμένη και σύντομη ημερομηνία για την απόφαση από τον εκτελεστικό διευθυντή για το εάν ή όχι κάποια πράξη έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων. Ε, αυτό ε, μας δημιουργούσε δυσχέρες γιατί πολλές φορές πρέπει να μπορέσεις να κρίνεις αναλυτικά διάφορα στοιχεία και τελικά καταλήξαμε στην διατύπωση ότι ο εκτελεστικός διευθυντής θα πάρει σύντομα μία απόφαση. Χωρίς λοιπόν όμως συγκεκριμένη προθεσμία γιατί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη πόσο σοβαρά είναι και πόσο σοβαρέ είναι οι πράξεις που μπορεί να έχουν διαπραχθεί. Και κάτι άλλο που προέκυψε και στι τελευταίε συζητήσει Έχουμε μια οριζόντια προσέγγιση για τα κύρια άρθρα με βάση την πρότυπη συμφωνία. Αυτά λοιπόν και βεβαίω να απαντήσω αν έχετε ερωτήσει. Και θα συνεχίσω να σα ενημερώνω. Ευχαριστούμε πολύ, Σάιμον, για αυτή την εξωτική παρουσίαση. Δυστυχώ κανένας από τους σκιώδεις εισηγητές δεν βρίσκεται Λυπούμε. Θέλω όμως να δω κατά πόσον άλλοι συνάδελφοι θέλουν το λόγο. Η κυρία Σιπέλ. Μπεργίτ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστούμε για την επισκόπηση. Ήδη στην παρουσίασή σας Αναφέρατε ότι κάποιες φορές κάποια ζητήματα επανέρχονται διαρκώς. Όμως, από την άλλη, νομίζω ότι κάθε κατάσταση για τα σύνορα οποιασδήποτε χώρας είναι και διαφορετική. Θέλω λοιπόν να σχολιάσω δύο σημεία. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Σύνοριοφυλακή θα, θα διεξάγει τι δραστηριότητέ τη βάσει των οδηγιών των αρχών τη τρίτη χώρα. Η ερώτησή μου είναι τι γίνεται αν οι οδηγίε για συγκεκριμένε δράσει αντιφάσκουν με του ευρωπαϊκού νόμου και κανόνε. Τι συμβαίνει τότε. Απλώ για επαλήθευση ρωτώ. Και η άλλη μου ερώτηση είναι για το μηχανισμό προσφυγών. Οι μετανάστες που βρίσκονται στα σύνορα γνωρίζουν τα δικαιώματά τους γνωρίζουν ότι υπάρχει μηχανισμός προσφυγών, υπάρχει τρόπος να τους πληροφορούμε και οι οργανισμοί πολιτών ω τρίτα μέρη μπορούν να έχουν πρόσβαση στον μηχανισμό αυτό των προσφυγών, μπορούν να υποβάλουν εκ μέρου κάποιου προσφυγή εφόσον υπάρξει πρόβλημα τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ευχαριστούμε, Γιούντιθ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η όλη μου αίσθηση και οι απόψει μου για το θέμα τη Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή είναι γνωστέ. Δεν θα επεκταθώ. Δύο θέλω να σχολιάσω, δύο σημεία. Όταν πήγαμε στα σύνορα Βουλγαρίας-Τουρκίας ε, για να δούμε τι κάνει εκεί η Frontex, είδαμε ότι υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ της ευρωπαϊκής πλευράς με τη βουλγαρική συνοριοφυλακή και του Τούρκου. Μάλιστα, η, ευρωπαϊκή, η ευρωπαϊκή πλευρά ήταν πολύ καλά εξοπλισμένη με ειδικά ε, γυαλιά και γυαλιά. Και όταν βλέπαν από την τουρκική πλευρά να έρχονται από στενού δρόμου άνθρωποι προ του φράχτε, ξέραν τι να κάνουν. Αυτό ήταν λίγο τρομακτικό βέβαια, γιατί δεν ξέρουμε αν κάποιο προσπαθούσε να πάει στο φράχτη για να πηδήξει και να σωθεί από την Τουρκία ή απλώ πλησίαζε. Ε, και μάλιστα ρώτησα του Βούλγαρου αν μπορούν να διακρίνουν κατά πόσον οι άνθρωποι αυτοί είναι Τούρκοι που προσπαθούν να δραπετεύσουν από την Τουρκία ή άλλε εθνικότητε. Κανεί δεν μπορούσε να απαντήσει σε απόσταση χιλιόμετρων με τα κιάλια. Άρα βρήκα μια συνεργασία υπερβολικά στενή για, τη για τα δικά μου τα γούστα. Όμω ε, η Ευρωπαϊκή Συνοροφυλακή ε, πρέπει να βρίσκεται κατά τι δύο πλευρέ των συνόρων. Αυτό κάνει την ε, συνεργασία ίσω ομαλότερη. Ακούγεται ενδιαφέρον στη θεωρία. Στην πράξη όμω, πώ θα βεβαιωθούμε ότι αυτοί που πραγματικά προσπαθούν να διαφύγουν από μια χώρα δεν θα του σταματήσουν στα σύνορα επειδή είναι τόσο όμορφη συνεργασία μεταξύ των σύνοροφυλακών μα. Και η άλλη μου ερώτηση, μπορείτε να αναλύσετε το αίτημα της Βοσνίας Ερζεγοβίνης που ε, ουσιαστικά θέλουν τη βοήθειά μας για να ελέγχουν τα σύνορα με την ε, Σερβία και το, το Μαυροβούνιο, αν κατάλαβα καλά. Άκουσα τι είπατε ε, και είπα, είδα ότι έχετε θετική στάση προς το αίτημα. Άρα, αν οδεύσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, θα αναλάβουμε ένα ρόλο που έχουμε διαδραματίσει στη δεκαετία του 90 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Μπορεί να το είχαμε κάνει τότε, αλλά για άλλους λόγους, όχι για έλεγχο της μετανάστευσης και των ε, προσφύγων, ε, των ροών προσφύγων. Είχε να κάνει με τις συγκρούσεις στα Βαλκάνια και το τι επικράτησε μετά. Δεν είμαι βεβαία ότι θα μου άρεσε να αναλάβω ένα τέτοιο ρόλο πάλι μεταξύ των ε, χωρών στα Βαλκάνια. Θέλετε λοιπόν να μας εξηγήσετε γιατί νομίζετε ότι ε, έχουν υποβάλει αυτό το αίτημα, γιατί έχουν αυτή την επιθυμία και κατά πόσον θα απαντήσετε θετικά. Δεν λέω ότι έτσι θα γίνει, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι μια ε, πιθανότητα για το μέλλον. Ευχαριστώ Γιούντι Σάιμον. Ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσουμε την ερώτηση της ερωτήσης της κυρίας Σίπελ νομίζω σε κάποιες υπό κάποια έννοια μπορούμε να τις απαντήσουμε με το κοινό τίτλο πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δύο-τρεις οπτικές γωνίες. Ρωτήσατε τι γίνεται αν ένα μέλος ομάδας λάβει οδηγία από τις αρχές που στέλνουν τις οδηγίες, τις αρχές της χώρας που τον έχει στείλει. Και αυτοί οι κανόνε τυχαίνει να αντιφάσκουν με την ευρωπαϊκή νομοθεσία ή τέλο πάντων παραβιάζουν, ενδεχομένω να παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Εδώ υπάρχουν ε, συγκεκριμένε ρήτρε τη συμφωνία και λένε ότι τα μέλη των ομάδων κατά την ε, άσκηση των καθηκόντων τους ε, υποτίθεται ότι πρέπει να σέβονται απολύτω τι θεμελιώδει ελευθερίε και τα δικαιώματα. Και κατά δεύτερο λόγο, οι συμφωνίε που είναι κάπω σφαιρικέ, συμφωνίε ομπρέλε, ε, επιτρέπουν τη θεωρητική εκδίπλωση δυνάμεων, αλλά στην πραγματικότητα έχουν να κάνουν και με το επιχειρησιακό πρόγραμμα δράση. Μια από τι απαιτήσει λοιπόν για τα προγράμματα των επιχειρήσεων είναι ότι πρέπει να ορίζονται συγκεκριμένε διατάξει ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Μεταξύ των οποίων ε, και η προστασία των προσωπικών δεδομένων, α πούμε. Άρα και στι βασικέ συμφωνίε και στι επιμέρου τα επιχειρησιακά δηλαδή προγράμματα, όλα αυτά καλύπτονται. Και κάτι άλλο που έχει συμβεί, το έχουμε δει να συμβαίνει, ε, κάποια χώρα εταίρος μπορεί να παραβιάζει τα βασικά δικαιώματα. Τους κανόνες των προσωπικών δεδομένων ή τους κανόνες της μη επαναπροώθησης, ας πούμε. Αυτό φαίνεται να είναι μια τάση που διαρκώ επανέρχεται. Οι συμφωνίε λοιπόν προβλέπουν εκτελεστικό διευθυντή του οργανισμού να μπορεί να διακόψει, να αναστείλει τη δράση σε περίπτωση που διαπιστωθούν τέτοιε παραβιάσει επανειλημμένω. Επίση, ρωτήσατε τι γίνεται με το μηχανισμό των προσφυγών τι να σα πω τώρα. Δεν μπορώ να πω αν κάθε μετανάστη προσπαθεί απελπισμένο να διασχίσει τα σύνορα γνωρίζοντα τι συμβαίνει με το μηχανισμό των προσφυγών, αλλά μπορώ να σα πω ότι ναι, οι συμφωνίε επιβάλλουν και για τι δύο πλευρέ να αναλάβουν την υποχρέωση να θεσπίσουν μηχανισμό προσφυγών. Στην περίπτωση των Δυτικών Βαλκανίων και των εταίρων μα εκεί, στι περισσότερε περιπτώσει, Συνήθω είναι ο εθνικός διαμεσολαβητής, ο ombudsman ή ο αντίστοιχος θεσμό που αναλαμβάνει για λογαριασμό του οργανισμού. Δηλαδή, εάν καταγγελθεί από ε, μια προσφυγή από υπάλληλο των ε, ευρωπαϊκών υπηρεσιών, ο μηχανισμός πρέπει να υπάρχει και θα χρησιμοποιηθεί για να εξεταστεί μια τέτοια προσφυγή. Και υπάρχει και υπεύθυνο για τα θεμελιώδη δικαιώματα και το Συμβουλευτικό Φόρουμ που είναι πολύ δραστήριο, όπω ξέρετε. Για τα ερωτήματα τη κυρία Αρχεντίνη τώρα. Και το τι γίνεται στα σύνορα Βουλγαρία-Τουρκία. Εκεί τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Σήμερα, όσοι από τον οργανισμό μα έχουν πάει εκεί, δεν έχουν εκτελεστικέ αρμοδιότητε. Η συνεργασία που σήμερα υπάρχει είναι κυρίω μεταξύ η επιχειρησιακή μάλλον συνεργασία που είδατε είναι κυρίω μεταξύ Βουλγαρική συνοροφυλακή και τουρκική. Όσοι από εμά έχουν πάει εκεί, περισσότερο συμβουλευτικό ρόλο έχουν και υποστηρικτικό. Δεν έχουν αναλάβει την ίδια τη διαχείριση των σύνορων και τα καθήκοντα σύνοροφυλάκων. Πάντω, πρέπει να δούμε κατά πόσον οι χώρε με τι οποίε συνάπτουμε τέτοιε συμφωνίε έχουν ένα σχετικό σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν μπορούμε να συνάψουμε συμφωνία με τρίτη χώρα που θα μας ανησυχούσε το πώς αντιμετωπίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα εν γέννη για τη Βοσνία τώρα και να τα εξηγήσω λίγο. Ας δούμε τι συμβαίνει από την οπτική γωνία των Βοσνίων. Μας λένε ότι έχουμε σοβαρές πιέσεις ως Βοσνία, ιδίως τα σύνορά μας με την Κροατία, με μετανάστες που προσπαθούν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ταυτόχρονα ως Βοσνία και στα σύνορά μας με τη Σερβία έχουμε σοβαρές πιέσεις, γιατί κάποιοι προσπαθούν να περάσουν από τη Σερβία παρανόμως σε εμά, θέλοντας μετά να επιχειρήσουν μια κίνηση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που μας έλεγε η Βοσνία λοιπόν, ότι θα ήθελαν να στείλουμε Ευρωπαίους νεροφύλακες με εκτελεστικές αρμοδιότητες στα εξωτερικά τους σύνορα, που δεν είναι σύνορα κοινά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι θα ήταν μέρος μιας προσέγγισης που θα τους επέτρεπε να ελέγξουν οι ίδιοι καλύτερα τα σύνορά τους και να ξαναδούν την όλη διαχείριση των συνόρων του. Σήμερα η νομική βάση τη Ευρωπαϊκή Συνοροφυλακή, ο σχετικό κανονισμό, δεν το επιτρέπει αυτό. Όμω, με τι προτινόμενε αλλαγέ, αυτέ που προτάθηκαν ήδη το Σεπτέμβριο, λέμε και περιγράφουμε τι τις ε, προποθέσει υπό τι οποίε μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Φυσικά υπάρχει και ένα σεβασμό, ένα επίπεδο σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών στις τρίτε χώρες, αλλά σε αυτέ τι περιπτώσεις θα μπορούσε να γίνει ε, εκδίπλωση και αποστολή κάποιων υπαλλήλων και σε τρίτη χώρα. Αλλά από την πλευρά των Βοσνίων έχω κατανόηση για το αίτημά του. Για αυτού είναι μεγάλη δυσκολία και μην σα πω ότι μπορεί να είναι και μεγαλύτερη το σύνορο με τη Σερβία από ότι με την Κροατία. Μάλιστα, κάποια άλλη ερώτηση είναι ναι. σύντομα. Μπορείτε τότε να μας πείτε γιατί είναι ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει κάτι τέτοιο, γιατί εγώ από ό,τι καταλαβαίνω μετακινούμε τα σύνορά μας λίγο πιο κάτω σε μια χώρα σε μια τρίτη χώρα. Ε, κοιτάξτε, εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς, ε, ποιος είναι ο σκοπός δηλαδή αυτής της συμφωνίας. Αν θεωρεί ότι είναι να σφραγιστούν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το λογικό θα ήταν να είμαστε στα σύνορα Βοσνίας Κροατίας. Εάν όμως θεωρεί ότι οι συμφωνίες αυτές έχουν στόχο να στηρίξουν εταίρους ε, στις κοινέ προκλήσεις, και να συνεργαστούμε με αμοιβαίο σεβασμό και να μην προσπαθούμε μόνο να ρίξουμε τον διπλανό μας ε, τότε αυτό είναι το σωστό και αυτό θεωρώ και εγώ ότι ήταν η καταλληλότερη πολιτική επιλογή δεν θα έπρεπε να έχω δώσει αυτή την ερώτηση συνεχίζουμε βέβαια στην παράδοση έτσι, των αντιπαραθέσεων με την Κομισιόν ευχαριστώ Σάιμον ε, ευχαριστούμε και την ομάδα σου για την παρουσίαση. Ευχαριστώ Μπίργκιτ και Τζούντιθ για τις ερωτήσεις. Να σας πω, συνάδελφοι, ότι οι τρεις υπόλοιπε ε, συμφωνίες με Βοσνία, Μαυροβούνιο και Σερβία θα ανατεθούν στην επόμενη συνεδρία των συντονιστών. Σάιμον, σε ευχαριστούμε. Η επόμενη παρουσίαση θα είναι πιο ήρεμη. Συνάδελφοι, περνάμε τώρα στο σημείο 5 για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης. Όπως θα θυμάστε, στις 12 Ιουνίου η Κομισιόν δημοσίευσε μια πρόταση κανονισμού για την σύσταση του ταμείου αυτού, ένα από τα προγράμματα που έχουν προταθεί στο πλαίσιο του ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ. Η εισηγήτριά μας είναι η Μίρια Μιντάλη. Υπέβαλε σχέδιο έκθεσης ε, στις 27 ε, Νοεμβρίου. Προθεσμία για τροπολογίες ήταν η 11 Δεκεμβρίου. Είναι 541 τον αριθμό νομίζω. Πάντα λέω κάποιον αριθμό, πάντα είναι λάθος. Μάλλον 546 θα είναι τελικά. Πολλές, εν περιπτώσει. Οπότε, Μίριαμ, κάνε την παρουσίασή σου για τις τροπολογίες και μετά θα κάνουμε μια σύντομη συζήτηση. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας, καλημέρα συνάδελφοι. Θεωρώ ότι εδώ πέρα τονίζεται η ανάγκη για δράση όταν μιλάμε για την νόμιμη μεταναστεύση και θα ήθελα εδώ πέρα να ευχαριστήσω όλους τους ηγητές για το ενδιαφέρον. Χτες μόλις ε, είδαμε μια χώρα, την Μάλτα, όπου έγινε μια αποβίβαση ανθρώπων που δεν τους δέχτηκε ένα άλλο κράτος μέλος και λίγες μέρες πιο πριν η ίδια χώρα, η Μάλτα, καλωσόρισε άλλα 249 άτομα. Μία περίπτωση είναι αυτή. Γνωρίζουμε και άλλες περιπτώσεις που συνέβησαν το 2018. Και είμαι σίγουρο ότι δεν θα είναι η τελευταία περίπτωση. Η κατάσταση αυτή τονίζει την διαφορά που υπάρχει μεταξύ των κρατών μελών που θέλουν να σώζουν ανθρώπινες ζωές και άλλους που δεν θέλουν να επιδείξουν αλληλεγγύη ως ε, εισηγήτρια αισθάνομαι μια υποχρέωση να αναφερθώ σε αυτά τα γεγονότα και να πω ότι ως συνομοθέτες είναι ευθύνη και καθήκον μας ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πιέσουμε τα κράτη-μέλη να κάνουν περισσότερα. Να δείξουμε αλληλεγγύη έμπρακτη, όχι μόνο στα λόγια. Και σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να συζητήσουμε πώς θα διαχειριστούμε 10 εκατομμύρια ευρώ Δράτομαι όμως της ευκαιρίας να πω ότι το θέμα δεν είναι μόνο χρηματικό. Είναι και θέμα των σωστών πολιτικών. Οι λύσεις ε, που βρίσκονται ενώ ε, κινδυνεύουν ζωές στην Μεσόγειο δεν είναι λύσεις ε, πανευρωπαϊκές. Είναι λύσεις ad hoc που λαμβάνουν μεμονωμένα κράτη-μέλη. Και έρχομαι λοιπόν στην αρχή της αλληλεγγύης, μια αρχή που αναφέρεται στις συνθήκες, άρθρο 80 της ε, συνθήκης και καθορίζει την αρχή της αλληλεγγύης και του διαμερισμού των ευθυνών και το ότι έχει και οικονομικές ε, συνέπειες για τα κρατημέλη. Έχω περιλάβει λοιπόν το άρθρο 80 ως μία από τις νομικές βάσεις του Ταμείου και χαίρομαι για το ότι υπάρχει μία διακομματική συνένεση από αυτού καθώς ε, και άλλοι ε, εισηγητές έχουν καταθέσει παρόμοιες τροπολογίες. Και βεβαίως αυτό θα το τονίσουμε και στις διαπραγματεύσεις μας με το Συμβούλιο. Δεύτερον, φαίνεται πως υπάρχει στήριξη της ε, πλειοψηφίας έτσι ώστε το Ταμείο αυτό να συνεχίσει να έχει ως μια προτεραιότητά του την ένταξη και πολιτικές ομάδες έχουν καταθέσει σχετικές τροπολογίες. Βεβαίως υπάρχουν και οι επιστροφές στον τίτλο, αλλά νομίζω ότι όλοι θα σκεφτούμε τα όσα έχουμε πει ως Επιτροπή για τον τίτλο αυτού του Ταμείου σε σχέση με τον κανονισμό κοινών διατάξεων. Ζητήσαμε δηλαδή να διατηρηθεί ο ίδιος τίτλος Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης. Τρίτο και πιο περίπλοκο, το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει και αφορά την σχέση με τρίτες χώρες πολλές ε, τροπολογίες έχουν καταδεθεί σχετικά και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί ένας συμβασμός, μια μέση λύση, δηλαδή να χρησιμοποιείται πρώτα απ' όλα το Ταμείο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να επιτρέπει και μια κάποια ευελιξία για δαπάνες σε τρίτες χώρες, υπό τον όρο ότι οι δαπάνες αυτές είναι εντός ορίων. Μετά, έχουμε την αρχή της εταιρικής σχέσης ε, που έχουν αναφέρει πολλές πολιτικές ομάδες ε, στις ε, τροπολογίες τους και αναμένω τις περαιτέρω συζητήσεις με τους υπόλοιπους και οδησίδες. Πέμπτον, έχουμε σημειώσει και αρκετές τροπολογίες στο άρθρο 8 συγκεκριμένα στον προϋπολογισμό, καθώς κάποιες ομάδες θέλουν να συζητήσουν την κατανομή των κονδυλίων μεταξύ των εθνικών προγραμμάτων και του θεματικού μέσου. Εγώ θεώρησα ότι δεν θα έπρεπε να αλλάξω την προτινόμενη κατανομή της Κομισιόν, αλλά θέλω να ακούσω από τους ηγετές το σκεπτικό τους. Από την άλλη, μία από τις κύριες αλλαγές που επέφερα αφορά την εισαγωγή ελάχιστων ποσοστών για κάποιες από τους στόχους ε, του Ταμείου. Το έχουν στηρίξει αυτό κάποιες ομάδες και θα είναι σημαντικό τομέα συμβασμών. Επιπλέον θα πρέπει να βρεθεί ένα συμβασμό για μια ελάχιστη κατανομή για τοπικές και περιφερειακές αρχές ε, που εφαρμόζουν δράσεις ένταξης ε, και έχουμε καταθέσει σχετικά τροπολογίες. Επίσης, οι θέσεις συγκλίνουν για την ανάγκη μεγαλύτερης διαφάνειας, παρακολούθησης και αξιολόγησης και βεβαίως ε, βελτιωμένη λογοδοσία στο Κοινοβούλιο. Καθώς επίσης ε, αυξήθηκε και το ποσοστό το οποίο απαιτείται από τα κρατη για να λάβουν τα κονδύλια μετά τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση στο 30% και βέβαια μετά έχουμε τα παρατήματα όπου έχω υποβάλει και εγώ πολλές ε, πρωτοβουλίες και ελπίζω να μπορέσουν να τις στηρίξουν περισσότερες ομάδες. Ελπίζω λοιπόν όλοι τις επόμενες ε, εβδομάδες να με στηρίξουν στην σύγκρουση αυτή με το Συμβούλιο. Να ευχαριστήσω λοιπόν τους και οδησίγητες για το πραγματικό ενδιαφέρον τους και αναμένω την επόμενη συνεδρία των συντονιστών στο Στρασβούργο και ελπίζω να έχουμε μέχρι το, τις πρώτες ε, συμβιβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Τέλεια παρουσίαση. Α, συγγνώμη. Λοιπόν, Μύρια, με ευχαριστούμε. Περνάμε στους κοιόδης. Γερούν Λέναρς. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και την κυρία Ντάλη για την εργασία της για το θέμα αυτό μέχρι τώρα και ευχαριστώ γιατί θέλησε να μας συμπεριλάβει όλους. Συναντηθήκαμε επανειλημμένα και θα έχουμε και την επόμενη εβδομάδα την ε, πρώτη συνεδρίαση των ε, σκιωδών και θα εξετάσουμε οποιασδήποτε συμβαστικέ. Ευχαριστώ όλου του συναδέλφου για τι 700 τροπολογίε. Δείχνει πόσο μα ενδιαφέρει το θέμα αλλά και πόσο σημαντικό είναι. Σύμφωνο, όπως είπε και την προηγούμενη φορά η συγκήτρια, ότι η ουσιώδη, η γνήσια αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών είναι σημαντικό στοιχείο στην αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Και χαίρομαι ότι το να μπει η αλληλεγγύη και η σωστή κατανομή στους στόχους του Ταμείου είναι κάτι επί του οποίου συμφωνούν όλες οι ομάδες. Και συμφωνώ και με τη φρασολογία που έχει εισαγάγει να στηρίξουμε την μόνιμη μετανάστευση σύμφωνα με τις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες των κρατών μελών. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για ένα θετικό τρόπο αντιμετώπισης Τώρα για το όνομα του Ταμείου. Προτείνω να αλλάχθεί το όνομα. Από πλευρά ΕΛΚ προτείνω να βάλουμε και τη λέξη και Ταμείο Επιστροφών. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι οι επιστροφές είναι σημαντικό τμήμα και το λιγότερο ε, εμφανές τμήμα αυτής της πολιτικής. Γιατί λοιπόν να μην μπει και στο όνομα. Καταλαβαίνω ότι αυτό δημιουργεί δυσχέρειες σε κάποιε πολιτικέ ομάδες. Γι' αυτό και όπως είπα ήδη στην εισηγήτρια, νομίζω ότι έχω μια πολύ καλή συμβαστική πρόταση. Να προτείνουμε να αλλάχθει το όνομα του Ταμείου, το, το Ταμείο να ονομάζεται το Ταμείο Μύριαν δηλαδή να είναι το Ταμείο για τις επιστροφές, την αλληλεγγύη, την ένταξη και την υποδοχή για τις τρίτες χώρες. Βεβαίως θέλουμε να ελέγχεται αυστηρά η χρηματοδότηση των τρίτων χωρών. Δεν συμφωνούμε όμως με τροπολογίες που αποκλείουν εντελώς κάποιες τρίτες χώρες ή που περιορίζουν την χρηματοδότηση μόνο σε γειτονικές τρίτες χώρες. Ξέρετε ότι Εάν θέλουμε να επιτύχουμε ένα συγκεκριμένο στόχο στη μεταναστευτική πολιτική, πρέπει να συνεργαστούμε συχνά με πολλέ χώρε. Για παράδειγμα, με τι χώρε ε, και προέλευση αλλά και διέλευση των μεταναστών. Πρέπει λοιπόν να εργαστούμε με όλε αυτέ τι χώρε. Βεβαίω. Έχουμε και το μέσο για την ανάπτυξη των γειτόνων και τη διεθνή συνεργασία αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο τον Ντίτσι θα έχει αποτελέσματα τα επόμενα χρόνια. Οπότε δεν πρέπει να εξαιρέσουμε ευθύ εξ αρχή την, ε, την συνεργασία με διάφορε χώρε. Κάτι άλλο που το ανέφερα και την προηγούμενη φορά. Το ταμείο αυτό πρέπει να είναι ευέλικτο για να προσαρμόζεται στις ε, προκλήσεις. Δεν μπορούμε να στηρίξουμε την εισαγωγή ελαχίστων αναγκών χρηματοδότησης μεταξύ των διαφόρων στόχων. Πρέπει να είναι στοχευμένη η χρηματοδότηση με βάση τις ε, πραγματικές ανάγκες που μπορεί να αλλάξουν ανα πάσα στιγμή. Αυτά συνοπτικά, αλλά προσβλέπω στη σημερινή συζήτηση και στην πρώτη μας ε, συνεδρίαση των σχεδόν την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος. Πολύ αναλυτικά και πλήρη όλα αυτά. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο δεν είναι κάπως καταβατικός ο τίτλος του Ταμείου. Ναι, σίγουρα δεν είχατε την πρόθεση αυτή, αλλά θα δούμε. Και θα δούμε πώς θα αντιδράσει και η συγγήτρια από αυτού. Πάση περιπτώσει αυτή είναι η δική μου άποψη. Αλλά σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλή παρουσίαση. ECI, κυρία Βίνμπερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Ανταλή, την εισηγήτρια. Ο προπολογισμό του Ταμείου για τη μετανάστευση δείχνει ότι έχουμε πολλά διαδοτικά προβλήματα. Είναι σημαντικό να τα επιλύσουμε, ούτω ώστε να εγγυηθούμε κάποια σταθερότητα και καλές λύσεις και για τις δικές μας χώρες που εδώ και χρόνια υφίστανται ε, σημαντική μετανάστευση, πολύ άριθμη. Είναι σημαντικό να μην ενθαρρύνουμε περαιτέρω μετανάστευση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί μετανάστε που έρχονται το κάνουν για οικονομικούς λόγους. Με διάφορα ανθρωπιστικά προσχήματα. Είναι σημαντικό το σύστημά μας λοιπόν να λειτουργεί πολύ καλά. Ο προπολογισμό μα λοιπόν πρέπει να ασχοληθεί με τους ε, γνήσιους ε, του άσυλο. Πρέπει να γίνεται σωστά ο διαχωρισμός μεταξύ αυτών και των οικονομικών μεταναστών. Και αυτοί οι οικονομικοί μετανάστες πρέπει να υπάρχει δυνατότητα συντόμως και αξιοπρεπώς να επιστραφούν. Αυτό είναι σημαντικό για την ε, κοινωνία των χωρών μας. Υπάρχουν ελλείψεις αυτά που προτείνονται. Λέμε ότι πρέπει να ενταχθούν οι μετανάστες. Δηλαδή εμείς θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Εμείς θα πρέπει να προσαρμόσουμε την κουλτούρα μας και τον πολιτισμό μας σε αυτή των ε, μεταναστών. Η κοινωνία μας πρέπει να προσαρμοστεί. Όχι. Τα άτομα αυτά που φτάνουν πρέπει να προσαρμοστούν στις κοινωνίες μας. Γι' αυτό το λόγο ο προπολογισμό μας του ταμείου αυτού προβλέπει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τις περιπτώσεις όπου μας εξαπατούν. Έρχονται δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό να μείνουν για οικονομικούς λόγους. Άρα αυτό που είναι αναγκαίο είναι να αποθαρρύνουμε τους οικονομικούς μετανάστες, να τους αποτρέψουμε. Αυτό είναι σημαντικό για την ευημερία και την ασφάλεια των συμπολιτών μας. Ευχαριστώ πολύ. Άλντε και Γκούε δεν βλέπω. Η Σκά Κέλλερ είναι η συντονίστρια των Πρασίνων. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την εργασία της και για το ότι μας ενημερώνει για όσα συμβαίνουν. Νομίζω ε, είναι πολύ περίεργο που η ένταξη απαλήφθηκε από τον τίτλο. Τώρα η Κομισιόν λέει ότι δεν χρειάζεται, δεν αλλάζει τίποτα. Αυτό με κάνει καχύποπτη. Πρέπει οπωσδήποτε να μπει η ένταξη. Και είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπιστεί η ανισορροπία της πρότασης της Κομισιόν. Ε, βάζει πολλά χρήματα στις επιστροφές. Αν δείτε το αμύφ και τι πρέπει να γίνει τι πρέπει να δώσουμε παντού στην Ευρώπη, σε διάφορες κοινότητες για να βοηθήσουμε την ένταξη. Έτσι μπορούμε να επιτύχουμε ουσιώδη πρόοδο. Και να προωθήσουμε και την ένταξη και την νόμιμη μετανάστευση. Υπάρχουν δυνατότητες, αλλά δεν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση. Αυτό πρέπει να κάνει το κατά τη γνώμη μας. Γι' αυτό υποβάλαμε τροπολογίες και βεβαίω προσβλέπουμε στην περαιτέρω συνεργασία με τους άλλους σκιώδε και την εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ Σκά. Θέλει κανεί άλλο το λόγο. Όχι, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Να επιστρέψω στην εισηγήτρια για το κλείσιμο. Ευχαριστώ πολύ. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Α, η πρώτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύντομα παρακαλώ. Σύντομα σα ξέχασα. Και μετά η Μίριαμ. Συγγνώμη. να κάνω μια μικρή διόρθωση γιατί υπάρχει κάποια παρανόηση για το ότι ίσως υπάρχει κάποια παρανόηση λοιπόν έλεγα το παράρτημα 1 που έχει την κλίδα κατανομής δεν λέει υποχρεωτικά που θα πάει χρηματοδότηση η πρότασή μας είναι ότι η χρηματοδότηση πρέπει να αντιμετωπίζει τις συγκεκριμένες ανάγκες των ε, διαφόρων κρατών μελών που μπορούν να διαφέρουν. Μπορεί να διαφέρουν. Το να λέγεται ότι δίνουμε προτεραιότητα στις επιστροφές ή ότι πολλά χρήματα πάνε στις επιστροφές δεν είναι κατά ανάγκη σωστό. Αυτή η κλίδα κατανομής αναφέρει τα κριτήρια βάσει των οποίων θα διανεμηθεί η χρηματοδότηση στα κράτη-μέλη. Δεν ειναι κατα αναγκη σωστο αυτη η κλιδα κατανομης αναφερει τα κριτηρια βαση των οποιων θα διανεμηθει η χρηματοδοτηση στα κρατη μελη δεν διευκρινιζει πώς ακριβώς θα δαπανηθούν. Δίνει τις εθνικές χρηματοδοτήσεις. Τα κράτη-μέλη φυσικά μπορούν να διοχετεύσουν τη χρηματοδότηση ανάλογα με τις ανάγκες τους. Τώρα για τον τίτλο του ταμείου. Δεν υπάρχει καμία κακή πρόθεση. Όπως ξέρετε έχουμε το πλήρες πακέτο του ΠΔΛΤΑΜΗ όπου θέλουμε η ένταξη να αντιμετωπιστεί γενικότερα, με πιο ευρύ τρόπο. Και επίσης και στο Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ, ESF ΣΥΝ. Επειδή λοιπόν αυτή η ένταξη των προσφύγων δεν είναι μόνο θέμα ασύλου και μετανάστευσης. Δεν χρειάζεται να αναφέρεται μόνο σε αυτό το ταμείο. Θέλουμε και τα δύο ταμεία να μπορούν να ασχοληθούν με αυτή την ένταξη για να μπορούν να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότησή τους τα κράτη-μέλη ανάλογα με τις ανάγκες τους. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Δεν κατάλαβα τι ακριβώς ε, εννοείται, αλλά ίσως καταλάβω μετά την παρέμβαση της συζήτριας. Κατάλαβα την πρώτη σας εξήγηση, αλλά όχι τη δεύτερη, αλλά βάση τόσο περιπτώσει η συγγήτρια. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους Κιώδης και την Επιτροπή. Συζητήσαμε μακρόν με την Επιτροπή για αυτό τον συγκεκριμένο κανονισμό και το συγκεκριμένο ταμείο και το συγκεκριμένο σημείο. Εγώ ως εισηγήτρια σε αυτή τη φάση δεν θεωρώ ότι επειδή είναι οριζόντιο στοιχείο η ένταξη δεν χρειάζεται να μην δώσουμε περισσότερη έμφαση σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, όπως είπαμε από την αρχή, το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα επίμαχο. Ξέρω ότι θα εκφραστούν πολύ διαφορετικές απόψεις. Αλλά η δουλειά μου είναι να καταλήξουμε σε βάσιμους συμβιβασμούς που να, μπορεί, που να μπορούν να συγκεντρώσουν πλειοψηφίες και στην Επιτροπή μας, στο Κοινοβούλιο. Αλλά ξέρω ότι κάποιες πολιτικές ομάδες ε, έχουν απόλυτη αντίθεση με κάποια σημεία. Αλλά κάποιες άλλες πολιτικές ομάδες νομίζω ότι μπορούν να βοηθήσουν να υπάρξει σύγκληση. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι γνήσια επιθυμώ να υπάρξει νομοθεσία που θα καλύπτει όλα τα σημεία που πρέπει να καλύπτονται. Ευχαριστώ τον κύριο Λένερς για τις προτάσεις τους για την ε, πρόταση το ταμείο αυτό να λέγεται Ταμείο Μύριαμ αλλά κοιτάξτε δεν είμαι τόσο ματαιόδοξη. Αλλά θέλω να ε, ε, υπενθυμίσω ότι σε ένα άλλο πλαίσιο ο εισηγητή του ΕΛΚ είχε προτείνει να λέγεται ΆΜΙΦ και όχι AMF αυτό το ταμείο. Εντάξει, καλά μπορούμε να δούμε τον τίτλο τελικά λέει ο πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ για τη σκληρή εργασία σας για αυτό το θέμα και ευχαριστώ και τους Κιώδης. Ωραία λοιπόν. Η ψηφοφορία ελπίζουμε 29 Ιανουαρίου να γίνει και ευχαριστώ την εισηγήτρια και τους κοιόδης και την Επιτροπή. Συνάδελφοι, τώρα να περάσουμε στο σημείο 6, Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Και πάλι εδώ έχουμε να εξετάσουμε τις τροπολογίες του θέματος. Η συγγετριά μας είναι η κυρία Μετσόλα. Η πρόταση τροπολογήθηκε περίπου 1600 φορές. Ευθύ αμέσω λοιπόν να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια για να μας παρουσιάσει το θέμα. Ευχαριστώ. Καλημέρα, Κλοντ. Είχαμε πολύ επικοδομητικές συζητήσεις τις προηγούμενες μέρες και εβδομάδες για την έκθεση αυτή μετά την παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης σε αυτή την Επιτροπή τον Νοέμβριο και πλην των τροπολογιών που υπέβαλε εγώ η Δία, λάβαμε 1.500 τροπολογίε συναδέλφων από αυτήν την Επιτροπή και από άλλε στην αρχική πρόταση τη Επιτροπή για έναν κανονισμό σε σχέση περί του Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακή. Όλοι ενδιαφέρθηκαν ε, πάρα πολύ από όλε τι πολιτικέ ομάδε, όλοι οι σκιώδει εισηγητέ και παρακολουθούν στενά τη διαδικασία. Δεν μείναμε αδρανείς Ήδη έχουμε επεξεργαστεί συμβαστικές λύσεις σε τεχνικό και πολιτικό επίπεδο. Ούτως ή άλλως δεν έχουμε και πολύ χρόνο σε αυτή τη θητεία. Θέλουμε λοιπόν να βιαστούμε για να ολοκληρωθεί το θέμα στο δυνατόν γρηγορότερα. Θεωρείται ένα θέμα προτεραιότητας για το Ευρωκοινοβούλιο και προφανώς αυτή της μεταχείρισης την χάνει και από εμάς τους ίδιους. Τα βασικά θέματα που θα μας απασχολήσουν στις διαπραγματεύσεις επί του θέματος είναι και αυτά που συγκέντρωσαν τις περισσότερες τροπολογίες. Η μεγαλύτερη δυσκολία από αυτά που προτείνει η Επιτροπή είναι το σώμα. Ε, το σώμα που θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτιστεί και οι σχετικέ τροπολογίε. Είναι σαφέ ότι το πρόγραμμα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ολοκληρωθεί η δημιουργία του σώματο ω το 2020 είναι ένα πρόβλημα και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Τροπολογίε λάβαμε και για τη σύνθεση του μόνιμου σώματο. Θέλουμε να υπάρχει διαλεκτικότητα για τη σύνθεση του και ταυτόχρονα να καλύπτονται οι ανάγκες του οργανισμού. Η πρόταση να, να προσθεθεί τέταρτη κατηγορία στο σώμα ένα ε, πουλ γρήγορη αντίδραση είναι κάτι που θέλουμε να λειτουργεί καλύτερα από ό,τι σήμερα και να μπορεί και να εκτυπλωθεί άμεσα. Έτσι μόνο θα πετύχουμε τους στόχους μας. Επίσης, πρέπει περισσότερες αρμοδιότητες να ανατεθούν σε αυτό το σώμα με περισσότερες αποσπάσεις βραχυπρόθεσμες ε, και άμεσες εφόσον χρειάζεται, για να μην υπάρχει αποστράγγιση των ε, ανθρώπινων πόρων, ιδιαίτερα των μικρών κρατών μελών ως προς την εκπαίδευση για τους μόνιμους αξιωματικούς του σώματος, και το κατά πόσο θα γίνεται απόσπαση μακροπρόθεσμη σύντομη, δηλαδή ή διαρκεία. Υπάρχουν πολλέ τροπολογίε εδώ από την ε, διαρκή εκπαίδευση ω προ την ε, Κεντρική Ευρωπαϊκή Ακαδημία για Συνοριοφύλακε που θα πρέπει να δημιουργηθεί. Θα πρέπει να εντοπίσουμε εδώ τι ακριβώ μα χρειάζεται. Πάντω, οι φιλοδοξότερε προτάσει είναι αυτέ που έχουν και μεγαλύτερο οικονομικό κόστο και ε, επηρεάζουν ε, το τι πόρους έχουν και τα κάτι μέλη ως προς τους εκπαιδευτές. Πρέπει να ε, βεβαιωθούμε ότι η επικουρικότητα και οι αρμοδιότητες των κρατών μελών ε, γίνονται σεβαστές. Οι σχετικές λοιπόν εδώ τροπολογίες συνδέουν τις δυνατότητες του οργανισμού να αναλάβει αποφάσεις μετά από συμφωνία με τα κράτη-μέλη και τη συνένεσή του. Άλλε τροπολογίε περιορίζουν τι εκτελεστικέ αρμοδιότητε των μόνιμων υπαλλήλων του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει εδώ να προβλεφθούν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε οι εκτελεστικές αρμοδιότητες που θα ανατεθούν να είναι μόνο οι αναγκαίες. Το Ευρωκοινοβούλιο ως προς το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, θέλει να το διασφαλίσει αυτό σε όλες τις θεμελιώδεις ε, σε όλες τις βασικές συμφωνίες. Με τις ε, τροπολογίες των σκιωδών λοιπόν κοιτάζουμε ε, η ρήτρα αυτή να ισχύει για όλο το σώμα του κειμένου. Άλλοι εισηγητές ε, δεν θέλουν να τα αφήσουμε αυτά και να μην επαναληφθεί η περίπτωση του ECBG του 2016. Εδώ υπάρχουν τροπολογίες σε πολλά σημεία του κειμένου. Όπω είπα προηγουμένω στου ε, θα πρέπει να υπάρξουν καλύτεροι ορισμοί για να αποφασίσουμε σωστά για το αν θα διατηρήσουμε αυτέ τι αναφορέ στα κέντρα ελέγχου, αν θα πρέπει να τροποποιήσουμε τον ορισμό του με κάποιο τρόπο, αν πρέπει να τα ε, αναφέρουμε μαζί με τα hotspot ή να τα καταργήσουμε όλα αυτά. Τέλος, η τελευταία παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι το κατά πόσο θα ασχολείται ο οργανισμός με τις επιστροφές σε τρίτες χώρες. Δεν θα ήθελα να ρισκάρω ο οργανισμός να παίρνει μέρος σε δραστηριότητες που ποτέ δεν επιτράπει εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, γι' αυτό ε, πρότεινα πέντε ρήτρε διασφάλιση στο σχέδιο εκθεσή μου, οι οποίε ενισχύθηκαν από αρκετέ τροπολογίε και προσθέτει λεπτομερέστερε διατάξει για τι σχετικέ διασφαλίσει των επιστροφών. Εδώ θα είμαστε αυστηρότατε στη διατύπωση. Η κατάσταση βεβαίω διαφέρει από το τι ίσχυε προδιετίες. Ιδίω επειδή υπάρχουν αρκετέ βασικέ συμφωνίε που έχουν συναυθεί μεταξύ του οργανισμού και αρκετών ε, μωρών χωρών. Θεωρώ ότι οι διατάξει αυτέ είναι μη διαπραγματεύσιμε και ο μόνο τρόπο που μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι η διαδικασία των επιστροφών γίνεται με σεβασμό των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι αυτό. Καταλαβαίνω βεβαίω ότι κάποιοι συνάδελφοι ανησυχούν ω προ αυτά, όμω είμαι πεπισμένοι ότι μπορούμε να επιδιώξουμε κάποια λύση σωστά εξισορροπημένη. Και πάλι, αν υπομονώ να ακούσω τα σχόλια των συναδέλφων και θα συνεχίσω να εργάζομαι άπνα με ε, τη συνεργασία των σκιωδών και των συνεργατών μας για να καταλήξουμε σε σωστές συμβαστικές λύσεις που θα γίνουν, αφού ε, όλα πάνε καλά, αποδεκτές από την απόλυτη πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Είναι ένα σημαντικό θέμα. Ε, θα περάσει στις 24 Ιανουαρίου σε ψηφοφορία να πάμε στο Σκιώδης. Μπίργκιτ, θες να πεις τίποτα από τους σοσιαλιστές. Όχι. Δεν είναι εδώ ο κύριος Νιντερμίλερ. Περνάμε στους εταιρικούς και μεταρρυθμιστές. Ο κύριος Βίστησεν. Κατά πρώτον, να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά της. Και κοιτάζοντα την πρόταση τη Επιτροπή, έχω πέντε σύντομε παρατηρήσει που θα προσπαθήσω να τι αναφέρω γιατί έχουν να κάνουν και με τη θέση μα ω ΙΣΙΑΡ. Πιστεύουμε λοιπόν στην ομάδα μα ότι είναι σημαντικό οργανισμό αυτό για την εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε. Μπορούμε να στηρίξουμε το συνολικό ε, το σκοπό της ανταλλαγής για να μην υπάρξει επιπλέον επάνθρωση. Επίσης, η σταδιακή αύξηση σε ανθρώπινους πόρους που προτείνει η συγγήτρια δεν είναι παράλογη για να μην αποσταγιστούν οι πόροι των κρατών μελών, οπότε και εδώ από την ομάδα μας μπορούμε να σας στηρίξουμε. Έπειτα βλέπω ότι υπάρχουν πολλές τροπολογίες για τη συγκεκριμένη εκπαίδευση των φυλάκων, όπως είπατε η συγγήτρια. Στου συντηρητικού και μεταρρυθμιστέ πιστεύουμε ότι ο καλύτερο τρόπο είναι να συμφωνήσουμε κάποια ελάχιστα πρότυπα για τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση. Και η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κέντρου για την εκπαίδευση, ίσως από την πλευρά του κόστους, να μην είναι και καλύτερη ιδέα. Μπορεί να το κάνουμε κι αλλιώ. Μετά δεν έχουμε αντίρρηση ως προς τις αρμοδιότητες επιστροφών που θα αναλάβει ο οργανισμός. Πολλές τροπολογίες βεβαίω δεν το θέλουν αυτό, είδαμε με τα λύπη μα. Όμω η συγκέντρια πιστεύουμε θα βρει τη σωστή ε, λύση και ένα κατάλληλο μοντέλο και για τις επιστροφές ώστε να διασφαλίζονται και τα ανθρώπινα δικαιώματα και να μην εγκαταλείψει πλήρω το πεδίο αυτοαρμοδιοτήτων οργανισμός, ε, ο οργανισμός εφόσον ήδη έχει κάποια σχετικά καθήκοντα. Επίσης υπάρχουν ανάμεικτα συναισθήματα ως προς το κατά πόσον ο οργανισμός μπορεί να προσφέρει συνδρομή σε τρίτες χώρες. Δεν είμαστε ακριβώς κατά τέτοιων αρμοδιοτήτων και της αναληψής τους, αλλά πρέπει να δούμε με ποια ακριβώς εντολή και σε τι πλαίσιο. Πάντως, είναι ευκαιρία για να ενισχύσουμε την ε, αξία και το νόημα της δουλειάς του οργανισμού αυτού. Και μια κόκκινη γραμμή για μας είναι το εξής. Εάν υπάρξει μετατόπιση στην πολιτική ηγεσία του οργανισμού, η ομάδα μας είναι πεπισμένη ότι θα υπάρξει πρόβλημα. Θα πρέπει την πολιτική ευθύνη να την έχουν τα κράτη-μέλη, όχι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα έπρεπε να έχει ζωτικό ρόλο στην καθοδήγηση και τον έλεγχο, τη διαχείριση του οργανισμού την ίδια. Πάντω πιστεύουμε ότι σε συνεργασία με του υπόλοιπου κοιότητε και την εισηγήτρια θα βρούμε καλέ συμβαστικέ λύσει. Ευχαριστούμε πολύ. Από την Άλντε, η κυρία Γκρισπέκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο κουβέντες είναι και η πρώτη συνεδρίαση της χρονιάς, οπότε καλή χρονιά. Για σας προσωπικώς κύριε Πρόεδρε και για όλους τους συνεργάτες, τους συναδέλφους και όσους δεν χαιρέτησα ακόμα, διαζώσεις αυτή τη σημαντική χρονιά. Να ευχαριστήσω την εισηγητριά μας, την Ρομπέρτα Μετσόλα, με τόσο σκληρή δουλειά, πραγματικά ε, κουραστική, και για ένα θέμα που είναι ιδιαίτερα προβεβλημένο για τους πολίτες που έχουν ευαισθησίες εδώ. Έχουμε ήδη προχωρήσει πολύ. Παρόλο που βρισκόμαστε σε σημείο λεπτό για να συμφωνήσουμε, αλλά οι αποκλήσεις απόψεων, χάρη στην δυνατότητα της ε, εισηγήτριας να μας ακούει και να βρίσκει συμβαστικές λύσεις, πιστεύουμε θα ξεπεραστεί. Οπότε μπορεί και να καταλήξουμε να έχουμε πια αυτό το εργαλείο για να καλύψουμε τις πραγματικές ανάγκες των Ευρωπαίων. Δύο λόγια για τις απόψεις της δικής μου, της κοινοβουλευτικής ομάδας. Από την δική μας πλευρά υποβάλαμε μια σειρά από τροπολογίες, διότι θέλουμε ισχυρότερη ευρωπαϊκή φιλοδοξία. Εδώ πολλές φορές αντίθετα στο ρεύμα αυτό έχουμε υποστηρίξει ανέκαθεν ως ομάδα και για την προστασία του χώρου Σέγγεν, πιο γενικά, και για την δημιουργία ενα τέτοιο εργαλείου σε ό,τι αφορά την προστασία των εξωτερικών συνόρων. Αυτό το σήμα κατά τεθέν, που είναι κατεξοχήν ευρωπαϊκό, το είχαμε πει και στο προηγούμενο ρίκαστ στην αναδιατύπωση που αφορούσε τον οργανισμό. Δύο-τρία λεπτομερέστερα σχόλια εντάχει. Πρώτα απ' όλα, σε σχέση με όσα είπαν οι προηγούμενοι για τη δημιουργία ενός μονίμου σώματος, εάν έχουμε ένα τέτοιο μόνιμο τάγμα, στράτευμα, σώμα ε, για την προστασία των συνόρων, σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε το πρόγραμμα που προτείνει αρχικώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι τελείω ανέφικτο. Θα πρέπει να βρούμε μια λύση για να μπορεί και να γίνει. Μην γίνουμε αντιπαραγωγικοί ούτε για το εργαλείο που θέλουμε να δημιουργήσουμε, ούτε για όσα περιμένουν από εμά οι Ευρωπαίοι. Και άλλα δυο σημαντικά για την ομάδα μα, αυτό το μόνιμο σώμα που θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκό, το συζητήσαμε και προηγουμένω, θα πρέπει. να αποτελείται κυρίως από μονίνους υπαλλήλους, την πρώτη κατηγορία που έχει προταθεί αυτή η ευρωπαϊκή κουλτούρα, αυτού του είδους η ενοποίηση δεν θα προχωρήσει, δεν θα γίνει πραγματικότητα εάν δεν ε, ακολουθήσουμε αυτήν την ε, επιλογή. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και τις σχετικές τροπολογίες για ένα κέντρο εκπαίδευσης ε, για το σώμα αυτό. Να υπάρξει μια κουλτούρα γύρω από την εκπαίδευση που να έχει ευρωπαϊκό περιεχόμενο. Αυτό θέλουμε να δημιουργηθεί στην πράξη και να λειτουργεί. Και μια δεύτερη παρατήρηση, έχουμε υποβάλει τροπολογίες για να επιμείνουμε στη διάσταση της προστασία των εξωτερικών συνόρων και την προστασία από το οργανωμένο έγκλημα. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν βεβαίως και με το πώς καταρτίζουμε τις μεταναστευτικέ μα πολιτικέ και τη διαδικασία των επιστροφών. Δεν θα είναι βεβαίω αυτό το κεντρικό ζήτημα των επιστροφών δηλαδή σε σχέση με τη δημιουργία του σώματο, αλλά πρέπει να επιμείνουμε και σε αυτό. Για τι επιστροφέ λοιπόν, Νομίζω πολλοί στις συζητήσεις που έγιναν ως τώρα υποστήριξαν ε, αφού εξέφρασαν τουλάχιστον την έκπληξή τους για το κατά πόσο μπορούμε να οργανώσουμε επιστροφές τρίτης χώρας προς τρίτη χώρα. Δεν είναι αυτός ο ρόλος του οργανισμού. Και πραγματικά ακόμα παραμένει η απορία μας, γιατί δεν έχουμε λάβει απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις νομικές της υπηρεσίες, για το πόσο, κατά πόσο μπορεί να συμπεριλαμβάνονται κέντρα ελέγχου. Τι θα πει κέντρα ελέγχου. Δεν υπάρχει ορισμός για τέτοιο πράγμα. Σε αντιδιαστολή με τα hot spot. Υπάρχει εδώ μια σχετική αμφισημία ε, για να μην το πω ε, μια γκρίζα ζώνη. Ελπίζω ότι βεβαίως αυτό το πέπλο μίχλης θα το διαλύσουμε με τις συζητήσεις μας αλλά θα είχε ενδιαφέρον η συγγήτρια να κατάφερε να τα καλύψει αυτά πολύ ε, ξεκάθαρα. Είμαι βέβαιο ότι θα το κάνει και το ίδιο και για την προστασία των δεδομένων. Αυτά ε, λίγο πολύ για να παρουσιάσω και τη θέση της ομάδας μου και βεβαίως σε αυτό το πνεύμα συνεργασίας θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις με την εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νάταλη. Από την ΚΟΕ δεν είναι εδώ κανείς. Δεν είναι εδώ η σιώδη συγγήτρια, δηλαδή. Οπότε θα μας τα πείσκα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Τονίσατε ήδη ποιες είναι οι τροπολογίες. Για εμάς δεν είναι τόσο σημαντικό το πόσες συνοριοφυλάκες υπάρχουν και τι κατηγορίες είναι. Μας ενδιαφέρει το τι κάνουν και πώς το κάνουν και αν κάνουν κάτι. Γιατί ήταν, ε, για μια τέτοια αύξηση ε, πρέπει να δούμε και ποιο είναι το πρόβλημα δηλαδή. Και συμφωνώ ότι πρέπει να παίξουν έναν ισχυρότερο ρόλο από ό,τι μέχρι τώρα στην καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος γιατί εκεί υπάρχει πρόβλημα που είναι κάτι το διαφορετικό από την μετανάστευση που ούτως ή άλλως ε, δεν μπορούν να σταματήσουν κάποιον να ζητήσει άσυλο. Από το ερώτημα είναι τι κάνουν και πώς θα το κάνουν. Συμφωνούμε με τη ρήτρα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πρέπει να αυξηθεί ο ρόλος της ε, Frontex ε, και η πτυχή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και βεβαίως της ε, αξιωματικού θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και συμφωνούμε με όλα τα ερωτηματικά για τα κέντρα ελέγχου και το πώς διαφέρουν από αυτά τα οποία ήδη υπάρχουν και το τι ακριβώς είναι. Και είμαστε επιφυλακτικοί αυτή τη στιγμή. Μέχρι να μας πείσετε, αλλά δεν το βλέπω. Και όσον αφορά τις επιστροφές, συμφωνούμε με τις ενισχύσεις της Νάταλη για το θέμα του να επιστρέψουμε κάποιον από τρίτη χώρα σε μια τέταρτη χώρα γιατί ό,τι ρήτρες και να έχουμε δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τι θα γίνει στη συνέχεια γιατί η Frontex θα δρά εκτός ε, της ε, δικαιοδοσίας της Ένωσης οπότε είμαστε πολύ αντίθετοι με αυτό κατά τα λοιπά περιμένουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία με τις κοινότητες εισηγητρίες σας ευχαριστώ το Ευχαριστώ, Κλοντ. Ευχαριστώ και εγώ την εισηγητρία, την κυρία Μετσόλα, για την δουλειά της. Δύσκολο το θέμα, επειδή δεν έχουμε και χρόνο και είναι και σημαντικό το θέμα και ιδιαίτερα προβεβλημένο. Έχουμε υποβάλει με τους συναδέλφους Κοράου και Καστάλντο 109 τροπολογίες επί της πρότασης της Επιτροπής τροπολογίες που θέλουν να ξεκαθαρίσουν ποιες είναι οι βασικές αρμοδιότητες του οργανισμού σε σχέση με τα όσα μπορούν να κάνουν και τα κράτη-μέλη. Διότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τους άντρες τους, ε, υποτίθεται, από, την, τον οργανισμό τα κράτη-μέλη ως υποστηρικτική δύναμη. Επίσης, Θέλουμε να δούμε κατά πόσον με την ε, αποτίμηση της κατάστασης της εξωτερική. σύνορα ενός μπορεί το κράτος μέλος, να, ο να αποφασίσει μόνος του τη συνδρομή. Επίσης θα πρέπει να δούμε τον έλεγχο που θα γίνεται στα σύνορα με βάση τις συστάσεις που θα προκύψουν από τα προηγούμενα και για το μόνιμο σώμα και την προστασία των συνόρων με 500 άντρε θα πρέπει να δούμε κατά πόσον θα είναι θελοντική η συμμετοχή εδώ των κρατών μελών. Η έδρα από την ε, Βαρσοβία στο Ρέτζο Καλάμπρια, στο νότο της Ιταλίας, έχει λογική. Είναι και αυτό μια πρότασή μας για σκοπούς ε, εγκύτητας και συνεργασίας στην περιοχή της Μεσογείου. Ζητήσαμε στήριξη του οργανισμού μόνο σε επίπεδο λογιστικό, διοικητικό και χωρίς παρεμβολή στις ε, καθήλυνα αρμοδιότητες, στις βασικές αρμοδιότητες των κρατών Και εν τέλει η δυνατότητα στα ελεγχόμενα όπως έχουν αναμονιστεί κέντρα να γίνεται και εξέταση αιτήσεων ασύλου είναι κάτι που δεν θέλουμε ώστε να μπορούν οι αιτούντες άσυλο να έρθουν στην επικράτεια του κράτους μέλους και να αρχίσουν να υποβάλουν αιτήσει ε, διεθνού προστασία. Αυτό είναι το περιεχόμενο των τροπολογιών μα και ευχαρίστω να συνεχίσουμε τι συζητήσει μα για να καταλήξουμε σε μια κοινή λύση για την εξέταση αυτού του τόσο σημαντικού θέματο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελειώσαμε λοιπόν με τους κοιόδης. Ποιος είναι? κύριος Λεοντίνη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να υπογραμμίσω πόσο σχολαστική στη δουλειά της και επιμελής ήταν η συνάδελφος Ματσόλα. Την ευχαριστούμε. Το θέμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Εκτοφυλακής είναι ζωτική σημασία, το γνωρίζουμε. Δεν θα μιλήσω συνολικά λοιπόν για το τι συναισθήματα μα προκαλεί η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάποιε προτάσει τροπολογιών τώρα, τι οποίε έχω βάλει εγώ ίδιες, ο ίδιο, μαζί με τη συνάδελφο Μουσολίνη και Ματέρα. Προτείνω η έδρα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού τη Ευρωπαϊκή Συνοφυλακή και Ακοτοφυλακή να πάει στην Κατάνια, στη Σικελία, καθώ Η πόλη αυτή βρίσκεται στο κέντρο τη Μεσογείου σε μια θέση στρατηγική για τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ κοντά στην Αφρική. Η Ιταλία είναι ένα από τα κράτη-μέλη που τα τελευταία χρόνια έχει προσφέρει τα περισσότερα προς την υποδοχή και τη διάσωση ζώων στη θάλασσα. Η επιλογή λοιπόν αυτή θα είχε και μεγάλη συμβολική αξία. Αυτή η πρόταση βεβαίως δεν πρέπει να κρυθεί ως απόρριψη της σημασίας της Βαρσοβίας και της Πολωνίας. Εκεί ας τους δώσουμε ένα ωραίο αντάλλαγμα. Αλλά είναι μια επιλογή που την επιβάλλουν τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πόλης της Κατάνιας, όπου βρίσκονται ήδη τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Task Force. Η περιοχή της Κατάνια έχει πάνω από 340.000 κατοίκους και η όλη η ευρύτερη περιοχή έχει το τρίτο αεροδρόμιο της Ιταλίας ως προς τις μετακινήσεις και τις αφήξεις. Είναι πολύ κοντά στην Βαλέτα που είναι έδρα της ΕΑΖΟ. Και αυτό θα επιτρέψει τη σύσφυξη των σχέσεων μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οργανισμών που ασχολούνται με τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης που ζούμε. Κατά τα άλλα, είμαι εντελώ στη διάθεσή σας να συζητήσουμε με την εισηγήτρια για να βρούμε ενδεχομένω μια πιο συγκεκριμένη πρόταση για το όλο θέμα. Ευχαριστώ. Να πω στην εισηγήτρια ότι έχουμε λίγο χρόνο. Οπότε δεν ξέρω αν μπορεί να μας πει κάτι η Προεδρία. Γιατί έχουμε κάποια ζητήματα στο Συμβούλιο αυτή τη στιγμή για τους 10.000. Δεν ξέρω, θέλετε να πείτε κάτι. Δύο λογάκια από την Κομισιόν ή η Προεδρία. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο. Μπορείτε να μας πείτε κάτι. Ωραία. Καλημέρα σε όλους. Προσωπώ την Προεδρία του Συμβουλίου από τη μόνιμη αντιπροσωπεία. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε τον λόγο. Να ευχαριστήσω και τα μέλη της Επιτροπής για την παρέμβασή τους και την θέση που έχουν στο πλαίσιο αυτού του φακέλου. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι αυτός ο φακέλος είναι πρώτη προτεραιότητα για την Προεδρία μας και έχοντας αυτό κατά νου εργαζόμαστε εντατικά στο Συμβούλιο για να βρούμε κάποιους συμβασμούς που θα αποδεχτούν τα περισσότερα κράτη-μέλη. Όπως ήδη γνωρίζετε η Αυστριακή Προεδρία κατέληξε σε μια γενική μερική προσέγγιση όσον αφορά τις επιστροφές και τη συνεργασία με τρίτες χώρες κατά το οποίο ακόμα συζητάτε για να βρείτε κάποιον συμβιβασμό ο στόχος μας είναι να καταλήξουμε σε μια διαπραγματευτική εντολή το συντομότερο δυνατόν και να ολοκληρώσουμε εντός της τρέχουσας Όσον αφορά το θέμα αυτό, προσπαθούμε να καταλήξουμε σε έναν συμβασμό στα εκκρεμή ζητήματα, δηλαδή τους 10.000 ή τις εκτελεστικές εξουσίες ε, και την κατανομή στα κράτη-μέλη. Και τις επόμενες εβδομάδες θα επικεντρωθούμε σε αυτά και ταυτόχρονα να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στα άλλα μέρη του κειμένου σκοπεύουν να είμαστε σε στενή επαφή με το Κοινοβούλιο και να προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε τον φάκελο αυτόν το συντομότερο να το ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ναι, όλοι αυτό θέλουν. Αλλά υπάρχουν κάποια πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα όπως οι 10.000. Είναι ενδιαφέρον ότι κάνετε την πρώτη παρέμβαση για την Προεδρία. Οι Υπουργοί έρχονται στις 23. Οπότε θα είναι αυτό ένα από τα ζητήματα. Και σας ευχαριστούμε που αναφέρατε ότι θέλετε να ενημερώνετε τους βουλευτές. Και αυτό πρέπει να γίνει για να τα καταφέρουμε εγκαίρως. Δεν ξέρω τώρα αν η συγγήτρια θέλει να ρωτήσει κάτι. Ναι, θέλω η Κομισιόν να απαντήσει στις ερωτήσεις των συναδέλφων, εάν γίνεται. Είστε έτοιμοι να απαντήσετε από την Κομισιόν. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Κοινοβουλίο, την εισηγήτρια και τους σκιώτες για τις ε, προσπάθειές τους Προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Κομισιόν να προχωρήσουμε το στομότερο δυνατόν. Όσον αφορά τον αριθμό των ερωτήσεων που ακούσαμε, προφανώς ε, έχουμε αρκετές ερωτήσεις. Η Κομισιόν, παραδείγματος χάρη, αναμένει να δει τις τροπολογίες και να τις αναλύσει όσον αφορά την επιβολή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και οπωσδήποτε θα περιμένουμε εδώ να δούμε ακριβώ αυτές τις ε, τροπολογίες όσον αφορά το μεγαλύτερο ρόλο στην καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος είναι και αυτό κάτι το πολύ ενδιαφέρον και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει σύγκρουση με τον άλλο ρόλο της Europol εδώ πέρα που θα πρέπει να υπάρχει η σωστή συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών τώρα να σχολιάσω ακριβώς αυτά τα δύο πράγματα ήθελα αυτή τη στιγμή και σας ευχαριστώ πάρα πολύ ωραία ευχαριστώ πάρα πολύ να ξαναρθούμε τώρα στην εισηγήτρια την κυρία Μετσόλα. Πόσο χρόνο έχω κύριε Πρόεδρε. Όσο θέλετε. Ε, καλά, μην το παρακάνετε, εντάξει. Προσέχετε τι μου λέτε, γιατί... Ε, εντάξει, είπαμε. Α, ευχαριστώ. Ε, σε κάποιους άλλους συναδέλφους δεν θα το έλεγα αυτό. Σας ευχαριστώ, Κλοντ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που εξέφρασαν την στήριξή τους στο έργο μου και την βούληση να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε κάποια ζητήματα. Έχουμε ίσως διαφορετικές ε, θέσεις, όμως θέλουμε να καταλήξουμε σε μια λύση στο θέμα αυτό. τα σχόλια που άκουσα από τους ε, συναδέλφους είναι ότι πράγματι το θέμα αυτό είναι ένα θέμα πρώτης προτεραιότητας ε, και πράγματι θέλουν να καταλήξουμε κατά τη διάρκεια αυτής της Προεδρίας. Θα ήθελα λοιπόν να επαναλάβω την προσήλωσή μας ε, ως Κοινοβούλιο στην συνεργασία με το Συμβούλιο και να επαναλάβω την ερώτησή μου θα ήθελα η Κομισιόν ε, να δει το σχόλιο για τα κέντρα ελέγχου και ε, επίσης ε, υπήρξε ένα θετικό σχόλιο στις προτάσεις μας για τα θεμελιώδη δικαιώματα και την υπηρεσία. Θα ήθελα επίσης να δούμε την πιθανότητα του να περιληφθεί στο κείμενο το τι εννοούμε όταν λέμε ότι η υπηρεσία πρέπει να έχει μεγαλύτερο ρόλο στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο είπε ο πρόσωπος της ε, Κομισιόν ότι πρέπει να δούμε και τους εκπροσώπους ε, των άλλων οργάνων πράγματι πρέπει ακριβώ να έχει ένα σχετικό ρόλο η υπηρεσία. Λοιπόν, τα σχόλια του ECR και των συντηρητικών για την εκπαίδευση. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει ε, στις συμβαστικές ε, προτάσεις μετά. για το σχολείο για τις επιστροφές ε, σε τρίτες ε, χώρες. Θα μπορούσαμε ίσως να ξεκαθαρίσουμε την συνεργασία με χώρες που έχουν ήδη κάποια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την υπηρεσία και στο πλαίσιο αυτό να περιλάβουμε και τροπολογίες ε, και πρόνοιες για τις επιστροφές. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε όμως ότι δεν αφαιρόμαστε σε σχέσεις με χώρες ε, με τις οποίες δεν έχουμε σχέση. Ε, οι, υπηρεσίες δεν έχουν κάποια σχέση. ομως σε ένα πλαίσιο, δηλαδή μιλάμε για χώρες με τις οποίες ήδη συνεργαζόμαστε και βλέπουμε τι είδους συνεργασία υπάρχει και τι θα μπορούσε να υπάρχει σε αυτόν τον τομέα. Εάν θέλει η χώρα να κάνει κάτι τέτοιο και αν τηρούνται όλοι οι κανόνες. Και, και η πατερμοσία για τους πρόσφυγες αν είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Ξέρω πως υπάρχουν διαφορετικές θέσεις αλλά θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στο θέμα αυτό των κέντρων ελέγχου και θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν να μου πει τι εννοούν ακριβώς εδώ πέρα και ποια είναι η νομική βάση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Όπως είπα, προσπαθούμε να έρθει αυτός 24 του μηνός αλλά είναι μεγάλο το θέμα. Ευχαριστώ λοιπόν τον την εισηγήτρια του Σκιώδη σε όλους τους συναδέλφους. Περνάμε τώρα στο σημείο 7. Κοινωτικός κώδικας θεωρήσεων. Έχουμε τον πρώτο τριμερή διάλογο που έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο. Συγητής είναι ο κύριος Λόπες Αγγιλάρ. Έχετε τον λόγο, Χουάν. Ευχαριστώ. Κλοντ, κύριε Πρόεδρε, για την ευκαιρία αυτή που μου δίνετε να ολοκληρώσουμε την ανταλλαγή απόψεων στο θέμα αυτό. Πρώτα απ' όλα να αναφερθώ σύντομα στα αποτελέσματα του πρώτου τριμερούς διαλόγου που έλαβε χώρα στις 13 Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο. Εκεί ξεκίνησε ο διάλογο με την Αυστριακή Προεδρία. για να καταλήξουμε σε αυτό το σημείο ξέρετε ότι εργαστήκαμε υπό πίεση δεν ήταν εύκολο για κανέναν ειδικά για το προσωπικό μας τώρα μας περιορίζουν βεβαίως οι νέες προθεσμίες που σχετίζονται με το ότι ε, πλησιάζουμε στο τέλος της ε, θητείας ε, θέλουμε να εγκριθεί ο κώδικας θεωρήσεων και πρέπει να καταληξούμε σε μια τελική συμφωνία στις 29 Ιανουαρίου και είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να υπάρξει η έγκριση από την Κορεπέρ στην 26 και να πάμε στην Λίμπε στις 27 ε, ή κάποια στιγμή τον Φεβρουάριο και να πάμε σε στην Ολομέλεια στην πρώτη ή δεύτερη Ολομέλεια του Μαρτίου αναλόγως. Οπότε θα πρέπει να εργαζόμαστε καθημερινά σε όλα τα επίπεδα. Οπότε θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστικοί και να προσπαθήσουμε να μείνουμε στη θέση της Ολομέλειας ε, του Δεκεμβρίου. Αυτό το μήνυμα πρέπει να στείλουμε στο Συμβουλίο αν θέλουμε να έχουμε επιτυχή ολοκλήρωση του τελωνιακού κώδικα σε αυτή την θητεία. Έχει φτάσει λοιπόν η ώρα των πράξεων της ευελιξίας ε, και του συμβιβασμού. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να περιορίσουμε στο ελάχιστο τις λεγόμενες κόκκινες γραμμές και να επιδείξουμε μια διαθεσιμότητα για ανταλλαγή απόψεων με το Συμβουλίο και να προσπαθήσουμε ακριβώς να βρούμε την ισορροπία στις διαπραγματεύσεις που έρχονται και τέλος είναι πρόφανες ότι είχαμε κάποιες ε, συναντήσεις, ολομέλειες, ε, σεμινάρια κτλ. με τους ενδιαφερόμενους ε, που έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους για τον κώδικα θεωρήσεων και προσπαθούμε ακριβώς ε, επιστήσουμε την προσοχή τους ε, στις διαπραγματεύσεις που λαμβάνουν χώρα και ακριβώς έχουν δείξει ότι πρόκειται για ένας δημαρχής. Αυτό ακριβώς ε, ελπίζουμε να έχουμε μια επιτυχία κατάληξη. Ο επόμενο τριμερή διάλογο θα γίνει στο Στρασβούργο στι 17 ε, του μηνό. Οπότε ελπίζω ότι ε, με τη συνεργασία των σκιωδών εισηγητών θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ. Κύριε Πέκερ, ο σκιώδη του ΕΛΚ. Θέλετε να πείτε κάτι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπα και χθες, στις συνεδρίες των εισηγητών, η οποία πήγε πολύ καλά, πολύ επικοδομητικά, σε μεγάλο βαθμό συμφωνούμε και κατανοούμε και τις διαφορετικότητες θέσεις, ε, των διαφορετικότητα των θέσεων των διαφοροπολικών πολιτικών ομάδων, αλλά υπάρχει ένα κείμενο που εγκρίθηκε από την Ολομέλεια, που μας υποχρεώνει, παρά τις διαφορετικές ε, απόψεις που μπορούμε να έχουμε, όπως για παράδειγμα, το θέμα ότι θέλουμε όχι μόνο κίνητρα, αλλά και κυρώσεις. Και γι' αυτό υποσχέθηκα στον εισηγητή ότι αυτός θα ηγηθεί των διαπραγματεύσεων και κάποιες ε, επιφυλάξεις που νομίζω ότι υπάρχουν στο Συμβούλιο δεν πρόκειται να τις αναφέρω και να τις προβάλλω. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πάνε πολύ επικοδομητικά τα πράγματα όπως το ανέφερε και ο εισηγητής μας μόλις τώρα. Ευχαριστώ κύριε Μπέκερ, λέει ο πρόεδρος. Άλντε. Ο κύριος Ντεπρέ. Ζερά, παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε μου. Ευχαριστώ και συγχαίρω τον εισηγητή μας, τον κύριο Λόπεθ Αγγιλάρ, για την ε, διαθεσιμότητά του και την καλή του διάθεση κατά τις συζητήσεις που κάναμε ως Σκιώδης. Στη χθεσινή συνεδρίαση τα πήγαμε πολύ καλά. Στηρίζουμε αποτελεσμα... Ε, αποφασιστικά την ανάγκη να γίνει ό,τι μπορεί να γίνει για να εγκριθεί αυτός ο κώδικας θεωρήσεων πριν το τέλος της ε, παρούσης κοινοβουλευτικής θητείας. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο πολιτικά αυτό για όλες τις πολιτικές ομάδες. Τώρα για το περιεχόμενο αυτών των συμφωνιών δεν έχουμε κόκκινες γραμμές που θα επέτρεπαν από πλευράς μας ε, τη συνένεση, αλλά εκφράσαμε σαφείς προτιμήσεις, τις οποίες γνωρίζει ο συγητής μας. Υπενθυμίζω για παράδειγμα ότι επιθυμούμε όλα τα κράτη-μέλη να κάνουν το αναγκαίο, ούτως ώστε να συνάψουν συμφωνίες με άλλα κράτη-μέλη για να εκπροσωπούνται όλοι προξενικά. Και όχι να αναθέτουμε αυτά τα καθήκοντα σε ιδιωτικές εταιρείες. Σαφώς προτιμούμε δημοσίους φορείς για αυτά τα θέματα. Τώρα για τα λεπτά θέματα, τις σχέσεις με την ε, επαναπρόθεση θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξουν επιπτώσεις για τα κράτη-μέλη που δεν συμφωνούν για την επανεισδοχή. Αλλά δεν πρέπει να πληρώνουν οι πολίτες. Θέλουμε οι ηγέτες των χωρών αυτών να υποστούν τις κυρώσεις. Αυτές είναι οι προτιμήσεις μας αλλά είμαστε ανοιχτοί σε συμβασμούς με το Συμβούλιο και εμπιστευόμεθα τον εισηγητή μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Ζερά, λέει ο πρόεδρος. Η Μαρή Κριστίν από πλευράς Γκουε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τον εισηγητή και το σύνολο των σκιωδών και όλους τους συνεργάτες μας που εργάζονται για το θέμα αυτό. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει γίνει πολλή δουλειά. Λυπάμαι που πρέπει ε, στα πλαίσια των πραγματεύσεων του Συμβούλιο να τελειώνουμε βεβιασμένα. Λόγω τέλους θητείας. Εντάξει, ας πούμε ότι το δεχόμεθα ως δικαιολογία. Υπενθυμίζω κάποιες κόκκινες γραμμές που έχουμε αλλά πρώτα απ' όλα υπενθυμίζω ότι ο κώδικας αυτός είναι μέσο που αφορά τα άτομα που θέλουν να παραμείνουν για ένα σύντομο χρονικό διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κυρίως οι τουρίστες και οι επιχειρηματίες. Όλοι οι περιορισμοί που θα αναφερθούν σε αυτό το κείμενο αφορούν τα εκατομμύρια θεωρήσεων που έρχονται ε, που χορηγούνται σε όλα αυτά τα άτομα που έρχονται κατά εκατομμύρια κάθε χρόνο. Και νομίζω λοιπόν ότι ορισμένες φορές ε, είναι λάθος μέσο για να αντιμετωπιστεί η λεγόμενη παράτυπη μετανάστευση. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Επειδή είμαστε μειοψηφία και η ομάδα μου και εγώ για τα θέματα αυτά, το σημειώνω επιμένω επιορισμένο. Συζητήσαμε, για παράδειγμα, το θέμα των εξαιρέσεων για τους ε, ανηλίκους και για όσους ε, διευκολύνουν τις πολιτιστικές, ε, σχολικές, πανεπιστημιακές ανταλλαγές και αθλητικές. Εντάξει, δεν αναφέρομαι στους φοιτητές που έρχονται εδώ για να σπουδάσουν στις χώρες μας, αλλά στους φοιτητές και πανεπιστημιακούς που έρχονται για επισκέψεις. Διαφωνούμε με το θέμα της σχέσης με την Συμφωνία Επανεσδοχής. Η θέση του κυρίου Ντεπρέ νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι ένας αποδεκτός συμβασμός. Δεν είναι δυνατόν οι πολίτες των χωρών αυτών να πληρώνουν τα σπασμένα των πολιτικών επανεισδοχής. Και επίσης, συμφωνώ με τον κύριο Ντεπρέ, όλο και περισσότερο και με ανισχύει βέβαια αυτό, συμφωνώ με τον κύριο Ντεπρέ <laughs> <laughs> Ναι, είναι πολύ ανησυχητικό, λέει ο πρόεδρο, αλλά συνεχίστε. Βεβαίω και συμφωνώ μαζί σα, κύριε Ντεπρέ. Με το τελευταίο που είπατε. Oui, exactement. Merci. αυτό ακριβώ, ναι. Για το θέμα. Κοιτάξτε, είναι τόσο σπάνιο να συμφωνούμε. Συμφωνώ λοιπόν ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στους, ε, σε δημόσιες υπηρεσίες για να χορηγούν θεωρήσεις. Γιατί ξέρουμε ότι όταν εμπλέκονται ιδιωτικές εταιρείες ανεβαίνει το κόστος. Πρέπει λοιπόν να ρυθμίζουμε εμείς το κόστος αν τελικά αναλαμβάνουν τις ε, βίζες ξένοι, ε, συγγνώμη, ιδιωτικές εταιρείες. Και συμφωνώ κύριε Ντεπρέ ότι πρέπει να παραμείνει η δυνατότητα χορήγησης βίζας στα σύνορα θα ήταν πολύ αρνητικό, ιδιαίτερα για τις περισσότερες θεωρήσεις, να καταργηθεί κάθε δυνατότητα χορήγησης θεωρήσεων στα σύνορα. Αυτές είναι οι κόκκινες γραμμές που ελπίζω λελογισμένα να σε αντιμετωπίσει το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Μαρή Χριστίνη, ο Πρόεδρος. Άννα, σύντομα παρακαλώ. Νομίζω ότι είναι μια φοβερή ε, δουλειά που έχουμε να κάνουμε πριν το τέλος της θητείας και για να δείξουμε πόσο σημαντική είναι η δουλειά μας ως κοινοβουλίου σε αυτήν ακριβώς τη θητεία. Πρέπει να το προβάλλουμε πολιτικώς αυτό το τελευταίο, αυτή την τελευταία μάχη του πολέμου που δίνουμε. Και πραγματικά νομίζω ότι το θέμα δεν είναι απλώς τεχνικό, δεν είναι γραφειοκρατικό. Ε, ε, αλλά πρόεδρε θα πρέπει να δώσουμε και σε εσά και στην Επιτροπο, Επιτροπή την δυνατότητα να επιφέρουμε ένα πλήγμα στο Συμβούλιο και να γίνει επιτέλους αυτό. Τι είναι αυτό που διακυβεύεται. Θέλουμε απλώς να ανακουφίσουμε την τεράστια καχυποψία κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτι που έληξε χθε με το Sea-Watch και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους με αυτές τις καταστάσεις που ε, αναγκάζουν τα κάτι μελη να λαμβάνουν τέτοιες αποφάσεις. Σε αποστολή στη Μελίγια είδαμε κόσμο Θυμάμαι μια οικογένεια Αιγυπτίων που τους είχαν χωρίσει στα σύνορα ε, έμποροι που τους είχαν εκβιάσει στα σύνορα του Μαρόκου να περά... και είχαν αφήσει την μητέρα με το μωρό να περάσουν και ο πατέρας με τα υπόλοιπα παιδιά μείναν από την άλλη πλευρά για να τους φέρουν και άλλα λεφτά. Και τέλος πάντων ε, τα πέρασαν όλα αυτά για να πάνε από την Αίγυπτο στη Μέλγία και δεν είχαν άλλο τρόπο, καμία νόμιμη οδό, καμιά ανθρωπιστική θεώρηση για να μπορέσουν ε, να διαφύγουν. για να πάνε από την Αίγυπτο Συριακή οικογένεια στη Μελίγια. Γι' αυτό λοιπόν αυτά που μας είπε ο Χουάν Φερνάντο και όλοι οι υπόλοιποι σκέωδεις που ασχολήθηκαν με το θέμα πρέπει να τους δώσουμε στήριξη. Χρειάζεται υποστήριξη για την δουλειά τους και τους ερχόμενους μήνες για τους τριμερείς. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ενημέρωση και υπογραμμίζω και πάλι αυτό που είπε στην αρχή. Αν θέλει αλλά πολύ σύντομα. Ευχαριστώ για τα σχόλια. Ήθελα απλώς να ενημερώσω για την κατάσταση πραγμάτων και για το ότι έχουμε πίεση χρόνου. Για την κατάσταση των πραγμάτων. Διότι έχουμε μόνο λίγες μέρες για να ολοκληρωθεί ο τριμερής διάλογος. Υπάρχει δυνατότητα να ολοκληρώσουμε με έγκριση το Μάρτιο στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ τους συνεργάτες μας, ευχαριστώ όλους τους κοιόδης και τα, τους άλλους συναδέλφους για τα σχόλιά τους και την Άννα που δεν είναι σκιώδης αλλά μόλις έκανε σχόλια. Ναι βεβαίως, βεβαίως ήταν σκληρή μάχη, σκληρή μάχη και πολύ παρατεταμένη. Χρόνια τώρα εργαζόμαστε για το θέμα αυτό, από τότε που υπήρξε η πρωτοβουλία της Κομισιόν. Και βεβαίω είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε συζητήσει όλα τα θέματα και από τεχνικής και πολιτικής άποψη ε, βίζες για ε, πολλαπλές εισόδους, σύστημα ε, αλληλουχίας που στηρίζεται από μερικά μεγάλα κράτη-μέλη και το θέμα της σύνδεσης με την επανεισδοχή. Αλλά καταλήξαμε σε μια λογική ισορροπία με βάση τους συμβασμούς που εγκρίναμε στην ψηφοφορία που κάναμε το Δεκέμβριο. Τώρα πρέπει να ολοκληρώσουμε την εργασία και σας ευχαριστώ για την καλή σας διάθεση, την ευελιξία σας για να επιτύχουμε συμβασμούς με το Συμβούλιο, ούτω ώστε να βελτιώσουμε την κατάσταση για το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη ότι ναι, Είναι πολύ σημαντική αυτή η άποψη που προτείναμε για την ανθρωπιστική βίζα να συμπληρώσουμε έτσι για τα περνοσμένα άτομα που διαφεύγουν μέσω της Μεσογείου το ε, οπλοστάσιο των δυνατοτήτων νόμιμης ε, εισόδου με βάση τις αρχές ε, τις οποίες υποτίθεται ότι εκπροσωπεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ και όλους τους συναδέλφους και να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Γιατί βλέπω ότι μπαίνει η εισηγήτρια. Γιατί το επόμενο θέμα λοιπόν είναι το 8 για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ε, Ευρωπαϊκών Υπευθύνων Σύνδεσης ε, Αναδιατύπωση. Υπευλήθησαν 177 τροπολογίες. Α, φεύγει η εισηγήτρια τώρα. Cecile, it's uh, report. Are Is okay? Α, τελικά δεν φεύγει. Καλά, μην τρέχεις, μην τρέχεις. Εντάξει. Ναι, ναι, τώρα έχουμε το θέμα σου. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Κάτσε με την ησυχία σου. Θα κάνω την παρουσίασή μου. Έτσι να υπογραμμίσω αυτό που είπε ο Χουάν Φερνάντο για το προσωπικό μα, Η Επιτροπή μας αυτή τη στιγμή έχει τους περισσότερους τριμερείς και θέλουμε να του ολοκληρώσουμε όλους ε, κατά τη διάρκεια της ε, Ρουμανικής Προεδρίας που θα είναι στην ουσία μόνο τρει ή τέσσερις μήνες ε, φοβερή δουλειά κάτι πρωτόγνωρο και για τα μέλη και για το προσωπικό μας καταπληκτική έχω και το κατάλογο αποτελεσμάτων αν από κάποια άλλη επιτροπή το αμφισβητήσει κανείς. Γι' αυτό οφείλεται στην εργασία σας και στην ποιότητά της. Σας ευχαριστώ που μας το υπενθυμίσατε. Σαφή όλα αυτά λοιπόν. Και νομίζω ότι δεν ζητήξαμε τι μπορούμε να κάνουμε. Να περάσουμε λοιπόν τώρα σε ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί, ένα περίπλοκο επίσης θέμα, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υπευθύνων Σύνδεσης για θέματα μετανάστευση. Λάβαμε 177 τροπολογίε. Η είναι η Κυριακή Έγκε, η οποία θα μα παρουσιάσει την άποψή τη επί των τροπολογιών. Εντάξει, παρακαλώ. Τι γνώμη σας λοιπόν επί των τροπολογιών επί της εκθέσεώς Ευχαριστώ Κλοντ. Και ε, επί τη ευκαιρία να ευχαριστήσω και τους κοιόδης εισηγητές για την συνεισφορά του στο σχέδιο έκθεσης. Όπως ε, ήδη ακούστηκε, έχουμε 177 τροπολογίες ε, που κατέθεσαν οι ομάδες και ήδη μας απασχολούν εδώ και κάποιες εβδομάδες στο τεχνικό επίπεδο. Πράγματι σκοπεύω να προτείνω στους κοιοδησηγητές ένα κοινό κείμενο που θα ανταποκρίνεται στις πρωτοβουλίες τους για να καταλήξουμε σε μια μορφή υπαλλήλου ο οποίος θα μπορεί να ασκεί αποτελεσματικά τις προτεραιότητες της Ένωσης στο πεδίο της μετανάστευσης. Ξεκινώντας από τα λιγότερο επίμαχα ζητήματα, θα πω το εξή. Υπάρχει μια μεγάλη σύγκληση των ομάδων, ειδικά όσον αφορά τον ορισμό του ε, υπαλλήλου αυτού συνδέσμου όσον αφορά τον ε, ρόλο του και τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχουν ακόμα κάποια ζητήματα που πρέπει να λυθούν όσον αφορά τις ε, λειτουργίες ε, αυτών των ανθρώπων. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε όμως κάτι το βασικό. Εάν από τη μία πλευρά είναι γεγονός πως οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι το alter ego των υπαλλήλων του ΟΗΕ που έχουν αποστολές ανθρωπιστικές σε τρίτε χώρε. Από την άλλη είναι επίση αλήθεια ότι δεν υποκαθιστούν τι δικαστικέ αρχές των κρατών μελών σε ζητήματα επαναπατρισμού όμω, ε, επαναλαμβάνουμε πω ε, στα πλαίσια των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων θα μπορούσαν να δώσουν πληροφορίες για την ανθρωπιστική κατάσταση των χωρών ε, φιλοξενίας και των κέντρων κρατήσεως. Και βεβαίω υπάρχει το άρθρο 3, παραγραφός 4, το οποίο προβλέπει ότι θα μπορούν να παρέχουν μια χρήσιμη στήριξη όχι μόνο στις ε, δραστηριότητες ε, επαναπατρισμού, αλλά και στις δραστηριότητες που αφορούν την καθοδήγηση και την συνοδεία των ατόμων που επαναπατρίζονται. Ε, βεβαίως είμαι ανοιχτή στην συνεννόηση με τους και συγητές ε, και στις διαπραγματεύσεις με την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Σεσίλ. Έχουμε μια σειρά από σκιώδη. Δεν ξέρω όμως αν είναι εδώ. Ναταλή, θες το λόγο. Mm. Ρομπέρτα, θε και εσύ. Ναι, ναι, έχω κάτι να πω, αλλά δεν πειράζει να προηγηθεί συνάδελφο. Όχι, όχι. Εσεί προηγήσετε απ' Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κυρία Μουσολίνη δεν μπορούσε να είναι σήμερα εδώ. Θεωρεί ότι οι υπάλληλοι, οι αξιωματικοί σύνδεσμοι, οι συνδετικοί αυτοί κρίκοι θα πρέπει να έχουν ε, σοβαρέ λειτουργίε, αλλά υπάρχει ο κίνδυνο οι λειτουργίες που αναλαμβάνουν στι χώρε προέλευση και διέλευση να επικαλύπτουν όσα κάνουν οι αρμόδιοι ευρωπαϊκοί οργανισμοί και αυτά θα πρέπει να τα αποφύγουμε. Υπ' αυτή την έννοια, οι τροπολογίε του ΕΛΚ σκοπό έχουν να επιδιώξουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι εθνικέ δυνάμει να διδραματίζουν ένα ρόλο συνεργασία με τι τρίτε χώρε για το θέμα τη μετανάστευση και με τρόπο αποτελεσματικό ώστε να μην υπάρξει και κατασπατάληση πόρων. Το ΕΛΚ ανέκαθεν επέμεινε στο ότι οι αξιωματικοί της μετανάστευσης θα πρέπει να προσφέρουν στήριξη στα θέματα επανεισδοχής και κρατήσεων. Γι' αυτό οι επαφές που έχουν με τις αρχές των τρίτων χωρών όπου έχουν ε, αποσταλεί θα πρέπει να αξιοποιηθούν για να μπορέσει να γίνει και η πολιτική επιστροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεσματικότερη. Ως ομάδα ε, θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι όσα ισχύουν για αυτού του υπαλλήλου προκύπτουν και από τα πρότυπα του ILO και τους υπόλοιπου υπαλλήλου της ευρωπαϊκή Ένωσης ώστε να, ενισχυθεί συμβολικά η ευρωπαϊκή αξία του ρόλου τους. Γι' αυτό το λόγο το ΕΛΚ έχει υποβάλει τροπολογίε που συνενώνει του τρει ορισμού του ΑΕΛΟ που έχει προτείνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει βεβαίω η αποστέλουσα αρχή να είναι αυτή που θα καθορίζει τα καθήκοντα και τι αρμοδιότητε των απολύων αυτών. Τέλο, η συγκεκριμένη μα πιστεύει ότι η περίοδο για την εξέταση του προγράμματο όπω θα εγκρίνεται από το Διευθυντικό Συμβούλιο θα πρέπει να μελετηθεί στα δύο χρόνια από τα τρία που την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θέλουμε μια ευρωπαϊκή απόκριση στη μετανάστευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κλείνοντα, να πω ότι το ΕΛΚ θα συνεχίσει να διαπραγματεύεται με επικοδομητικό τρόπο με του υπόλοιπου σκιώδου. Ευχαριστούμε, Ρομπέρτα. Από την Άλντε, η Ναταλή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σειρά μου να πω ότι και εμείς Χαιρόμαστε με την ε, πρόοδο στις συζητήσεις μας για τους αξιωματικούς αυτούς ε, διαδικτύωσης ή συνδέσμους και ευχαριστούμε και τη συνάδελφο Κιέγγε γιατί είναι δύσκολη η προσπάθειά της αλλά και επικοδομητική. Είναι λεπτό το θέμα. Έχουμε υποβάλει μια σειρά από τροπολογίες, θα συνεχίσουμε και θα τις εξετάσετε είμαι βεβαία και πολλές έχουν ήδη ενσωματωθεί στις συμβαστικές λύσεις. Η πρωταρχική στόχη για την ομάδα μας είναι να έχουμε μια θέση του Κοινοβουλίου που να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, μόλις υπόθηκε, τα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών και όλος ιδιαίτερος, και εδώ θέλω να επιμείνω, των ανηλίκων παιδιών είτε συνοδεύονται είτε όχι. Διότι έχουμε ευθύνη και απέναντί τους. Αυτά σε μεγάλο βαθμό καλύπτονται και από τις τροπολογίες, ιδίως για την προστασία των πλέον ε, ευάλωτων και εκτεθειμένων. Και δύο διευκρινήσεις Μιλάμε εδώ για διαφορετικά είδη υπαλλήλων συνδέσμων διαδικτύωση ε, στην αναδιατύπωση αυτή που θα αναλάβουν και αρμοδιότητες ανάλογα με την αρχική τους εκπαίδευση αλλά και ανάλογα με την πείρα τους. Πρέπει αυτό να το προσέξουμε. Ένας υπάλληλο που είναι από την αστυνομία μην πάει σε αποστολές που δεν έχουν καμία σχέση με τα αστυνομικά ή ασχοληθεί περισσότερο με την οικοδόμη από ότι με την ασφάλεια. Νομίζω θα τα καταφέρουμε παρόλα αυτά. Δεν θέλουμε να αρχίσουμε πάλι τα σεμινάρια εκπαίδευση ε, και να επαναλαμβάνουμε και άλλου κύκλου εκπαίδευση και άλλου, ιδίω αυτά που έχουν οργανωθεί με τον κύκλο μαθημάτων για το Ευρωπαϊκό Σώμα Ακτοφυλακή και αυτά που θα γίνουν και για το Σώμα του Αρσίλου. Θα τα δούμε βεβαίω λεπτομερέστερα. Έχουμε και άλλε συζητήσει στο πρόγραμμα και όπω είπε και η Σεσίλη είναι κάποια τεχνικά ζητήματα και πολιτικά τα οποία πρέπει ακόμη να πληθούν. Θα τα δούμε την ε, προσεχή εβδομάδα η ομάδα μου θα είναι διαρκώς ε, διαθέσιμη για να βρεθούν οι σωστές λύσεις για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Δεν σας πρόσεξα, γιατί δεν είστε στον κατάλογο των σχεδόν. Παρακαλώ, έχετε το λόγο από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Ευχαριστώ. Βεβαίως, θα υποστηρίξουμε όλες τις προσπάθειες για την αποτελεσματική προστασία των συνόρων μας και την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης. Εμείς στην ομάδα μας ανησυχούμε. Ανησυχούμε γιατί υπάρχουν κάποιες τροπολογίες που μας ενοχλούν. Χρησιμοποιούνται για να γίνει προώθηση της μετανάστευσης. Και μάλιστα με μία εκμετάλλευση της έννοιας της οικογενειακής επανένωσης. Άλλο τα δικαιώματα όσων ε, είναι μειονεκτούντες και άλλο διόγκωση της μετανάστευσης. Η διόγκωση της μετανάστευσης, οποιαδήποτε διόγκωση, θα κάνει τα κράτη-μέλη να αντιδράσουν ακόμα χειρότερα στους μετανάστες. Καλό θα ήταν λοιπόν να αποφύγουμε τέτοιες δράσεις που θα οδηγήσουν σε αυτή την κλιμάκωση της μετανάστευσης. Ε, μας ε, ενδιαφέρει πολύ αυτή η τροπολογία μας να περάσει. Διότι δεν μπορούμε να ενθαρρύνουμε τις χώρες να πάψουν να προστατεύουν τα σύνορά τους. Αυτό είναι επίθεση κατά του κάτους δικαίου. Τα σύνορα οφείλουμε να τα προστατεύουμε. Δεν μπορούμε να αποκύπτουμε στις πιέσεις. Οι χώρες να εγκαταλείπουν τα συνταγματικά τους δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Δεν θέλουμε αυτοί οι υπάλληλοι σύνδεσμοι να γίνουν εκπρόσωποι τύπου για τα θέματα μετανάστευσης και να υποκαταστήσουν ε, τους συνοριοφύλακες ας πούμε. Να υποστηρίξουν τα κράτη-μέλη, εντάξει, αλλά όχι να τους πάρουν ε, και τη δουλειά μας από τα χέρια ή να τους περιορίσουν στο τι μπορούν να κάνουν. Θα υποστηρίξουμε λοιπόν την έκθεση αυτή, αλλά μόνον εάν η θέση μας περάσει. Απλώς να σας θυμίσω ότι εδώ δεν υπάρχει πολιτική διαφωνία, ούτε πολιτικές επιλογές πρέπει να κάνουμε. Το ζητούμενο είναι να προστατεύσουμε τους πολίτε μας και να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο περιβάλλον που να επιτρέπει σε όσους είναι απαραίτητοι να περάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνον εφόσον υπάρχει λόγος. Ευχαριστούμε από την ΚΟΕ κυρία Βρεζιά. Καταρχάς και εγώ να ευχαριστήσω τη Σεσίλ. Έχει κάνει τρομερή δουλειά. Και πραγματικά και μένα με εκφράζει σε μεγάλο βαθμό με αυτά που προτείνει. Και με τις συμβαστικές της που νομίζω θα τις λάβουμε που να είναι. Σε κάποια σημεία διαφωνώ, ξέρω ότι δεν θα γίνει ακουστή άποψή μου, αλλά θέλω να τα πω. Καλό είναι να μην έχουμε ιδεολογικά κολλήματα σε σχέση με το θέμα της μετανάστευσης. Όλοι οι μετανάστες πρέπει να τη χάνουν της ίδιας μεταχείρισης. Με σοκάρει που μας κάνει κηρύγματα ένας Πολωνός βουλευτής για το θέμα αυτό, ενώ η Πολωνία είναι υπεύθυνη για το 60% των οικονομικών μεταναστών που μεταναστεύουν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μας τα κηρύγματα Πολωνία, αλλά η Πολωνία να είναι και συνεπής με αυτά που κάνει με τον εαυτό της και να ε, μην ξεχνάω ότι είναι η πρώτη χώρα που ε, στέλνει οικονομικούς μετανάστες. Μιλάμε για μετανάστευση υπό όλες τις έννοιες. Κύριε Γιούρεκ, άμα θέλετε να σας τους δείξω και να σας τους στείλω και πίσω τους Πολωνούς. Η μετανάστευση λοιπόν είναι ένα θέμα σφαιρικό, συνολικό δεν μιλάμε μόνο για τους άτυπους μετανάστες, για τους λάθρο μετανάστες. Πρέπει λοιπόν να ισχυθεί η διάστευση της πρόληψης, εντάξει, και η λαθρομετανάστευση να μην επιτρέπεται, να μην έχουμε καταστάσεις παράνομες και άτυπες, αλλά την νόμιμη μετανάστευση πρέπει κάπως να τη χειριστούμε. Αυτό τι σημαίνει λοιπόν. Ότι θα έχουμε και ανθρώπους που μεταναστεύουν εσωτερικώς και εξωτερικώς. Όχι μόνο αυτούς που έρχονται υποχρεωμένοι από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να κοιτάζουμε λοιπόν τις ροές και τις αυξητικές τάσεις. Ναι, υπάρχει Ήπειρος, από την οποία έχουμε περισσότερες ε, αφήξεις, 20% από την Ασία συγκεκριμένα, ε, λαθρομετανάστευσης. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τις ενόπλες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή. Έχουμε και Ινδούς και Κινέζους να σταματήσουμε λοιπόν να λέμε ότι μας κατέβει για το θέμα αυτό και να μην έχουμε μόνο ιδεολογικές παροπίδες. Ούτε να κάνουμε κηρύγματα στους υπόλοιπους γιατί αρχίζει να γίνεται λίγο κουραστικό. Ε, τώρα για τους υπαλλήλους συνδέσμους πιστεύω ότι πραγματικά ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι κάτι που θα πρέπει να πρετανεύσει. Ε, όλοι οι μετανάστε έχουν δικαιώματα και όλα τα κράτη-μέλη έχουν υποχρεώσει βάσει του διεθνού δικαίου. Καλό θα ήταν να υπάρχει μια ισορροπία προ το θέμα αυτό. Θα έπρεπε λοιπόν οι υπάλληλοι αυτοί, οι αξιωματικοί ε, διαδικτύωση να επιτρέπουν αυτό να διασφαλιστεί. Σε ένα πλαίσιο που μάλιστα γίνεται όλο και περισσότερο ασαφέ. Θα ήθελα όμω οι αξιωματικοί αυτοί για τη διαδικτύωση και νομίζω ότι και η Σεσίλ και η Ναταλή είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένε ω προ αυτό, να μην μετατραπούν σε πράκτορες της ασφάλειας το, για την, και της πολιτικής ασφάλειας. Στα πλαίσια της διεθνούς συνεργασίας μην γίνουν οι σωματοφύλακες για τα υπόλοιπα. Θα πρέπει να προσέξουμε λοιπόν το ρόλο αυτών των αξιωματικών, των υπαλλήλων διαδικτύωσης. Θα πρέπει να είναι ε, πολύ σωστά ε, καταρτισμένος για να μην προσπαθήσουμε απλώς να ξεφύγουμε από το θέμα της, μετανάστε... θέμα της μετανάστευσης από ένα παράδρομο. Όταν χαράζουμε νομοθεσία πρέπει να έχουμε ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Το θέμα της μετανάστευσης είναι ένα θέμα σφαιρικό, ε, συνολικό και έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Ευχαριστούμε, συνάδελφοι. Έχουμε φτάσει περίπου στο τέλος του χρόνου μας, έχουμε μέχρι τις 11, οπότε λίγο να επιταχύνουμε. Για το θέμα αυτό να ζητήσω από τη Σεσίλα να έχει να προσθέσει κάτι, να καταλήξει. Ευχαριστώ, Κλοντ. Ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους που τρόπον τηνά μπόρεσαν να στηρίξουν την όλη μας προσπάθεια. Πάρα πολλές τροπολογίες καλύφθηκαν. Όλες τις εξετάσαμε και να επαναλάβω, όπως και περισσότεροι συνάδελφοι, ότι συμφωνώ. Ε, πρέπει να αποφύγουμε να μετατρέψουμε αυτήν την προσπάθεια, τη δουλειά τους, υπαλλήλου διαδικτύωσης, σε ένα ζήτημα ιδεολογικού περιεχομένου. Να είμαστε πολύ πρακτικοί και να κοιτάξουμε να δώσουμε μια πραγματική απόκριση στο φαινόμενο της μετανάστευσης. Πρέπει να ανταποκριθούμε με τρόπο σφαιρικό και μια συνολική προσέγγιση. Ευχαριστώ πολύ για τη σκληρή σου δουλειά για το θέμα αυτό, Σεσίλ. Καλή τύχη σε όλους τους συναδέλφους γι' αυτό. Ξέρω ότι κάποιοι θέλουν να δευτερολογήσουν, αλλά δεν θα μπορέσω να το επιτρέψω, γιατί έχουμε 11 η ώρα της ψηφοφορίας και έχουμε και άλλο θέμα. Σας παρακαλώ λοιπόν δείξτε κατανόηση, σας ευχαριστώ. Ευτυχώς το επόμενο θέμα είναι δική μου η έκθεση. Το σημείο 9 κατάλογος τρίτων χωρών υπήρχοι των οποίων πρέπει να έχουν ε, βίζα στα εξωτερικά σύνορα και των οποίων έξερουν ε, ως αποτέλεσμα της ε, εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου. Η πρόταση αυτή της Κομισιόν είναι απαραίτητη στο πλαίσιο των ενεργειών του Brexit. Τι είναι αυτό, δεν το ξέρω από αυτό. Όσον αφορά ακριβώς ε, το τι θα γίνει με τους Βρετανούς πολίτες μετά το Brexit που θα πρέπει να εξαιρούνται από την απέτηση θεωρήσεων όταν ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για σύντομη διαμονή. Στο άρθρο 2 λέει ότι θα υπάρχει ένας ε, μηχανισμός αμοιβαιότητας σύμφωνα με τον κανονισμό 539-2001 στην περίπτωση στην οποία το Ηνωμένο Βασίλειο εισαγάγει απέτηση θεώρησης και θα ισχύσει από τις 30 ε, Μαρτίου 2019 στο πολύ, σύντομη, στο πολύ σύντομο σχέδιο εκθεσής προτείνω να δεχτούμε την πρόταση της Κομισιόν χωρίς τροπολογίες. Έχουμε κάποιους κοιόδης. Ε, ένας από αυτούς είναι εδώ. Κάποιο συνάδελφο λοιπόν θέλει να παρέμβει, παρακαλώ. η Μαρτίνα Άντρεσον είναι εδώ, η σκιώδης εισηγήτρια της Γκουε. Να ακούσουμε πρώτα την Μαρτίνα που είναι σκιώδη εισηγήτρια ο Ντάν είσαι και εσείς σκιώδης Μαρτίνα Συμφωνώ με την θέση σας. Οι Βρετανοί πολίτες ε, και από τη Βόρεια Ιρλανδία θα πρέπει να εξαίρονται από την Βίζα όταν ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για σύντομη διαμονή. Να σας πενθυμίσω την θέση που έχουμε λάβει για τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής και για να διασφαλιστεί στο σύνολό της για να μην υπάρχει καμία διαταραχή στο καθεστώς και το πλαίσιο στο οποίο εφαρμόζεται αυτή η συμφωνία οπότε πρέπει να εστιάσουμε ακριβώς στο να έχουμε κάποιες διευθετήσεις που θα αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες των ανθρώπων στη Βόρεια Ελλανδία όπως ξέρετε σύμφωνα με την συμφωνία αυτή δικαιούται αυτοί οι άνθρωποι βρετανική ή ιρλανδική υπηκότητα και αυτό έχει ε, καταγραφεί και στο Σύνταγμα της Ιρλανδίας οπότε μπορούν να θεωρηθούν Ιρλανδοί οπότε πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος στους Ιρλανδούς πολίτες που ζουν στη Βόρεια Ιρλανδία γιατί όταν μιλάμε για πολίτες της Ένωσης ε, που περιλαμβάνουν και τους Ιρλανδούς πολίτες στην ε, Βόρεια Ιρλανδία δεν θα πρέπει αυτοί να παγιδευτούν ε, στην συζήτησή μας οπότε θα πρέπει να ισχύουν τα συμφωνημένα για τη Βόρεια Ιρλανδία και θα συνεργαστώ μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ντάνταλτον. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ και εγώ. Αυτή είναι η μόνη λογική προσέγγιση που νομίζω θα καθισκάσει πολλέ ανησυχίε που υπάρχουν για την διαδικασία. Από την δική μας τη σκοπιά συμφωνούμε. Μια λογική προσέγγιση συμφωνούμε και με την Κομισιόν. Και το ίδιο συμβαίνει και στο Λονδίνο, σας διαβεβαιώ. Όπως είπαμε είναι και θέμα αμοιβαιότητας όπως πάντα σε αυτά τα ζητήματα και την ίδια άποψη και διαδικασία θα ακολουθήσουν και στο Λονδίνο. Να αναφερθώ στην ε, συνάδελφο που μόλις μίλησε βεβαίως η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής λέει πως δεν θα πρέπει να υπάρχουν και εμπόδια μεταξύ Βορείου Ιρλανδίας και Λονδίνου. Πρέπει και αυτό να το έχουμε κατά νου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ίσως ε, η Βουλή των Κοινοτήτων θα μπορούσε να παραδειγματιστεί από την δική μας την συνενετική συζήτηση για όλα τα ζητήματα. Βεβαίω αυτό δεν προδικάζει τίποτα για τα άλλα ζητήματα των Βρετανών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και τα θέματα αμοιβιότητας. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τη λογική σας προσέγγιση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τζιούρεκ, ε, για κάτι άλλο θέλετε να πείτε για το προηγούμενο θέμα. Πείτε μας. Σας ευχαριστώ. Όχι, ήθελα να επισημάνω το ότι ε, το δικαίωμα στην απάντηση όταν ε, αναφέρεται το όνομα ενός βουλευτή αναφέρεται στον κανονισμό. Αλλιώ δεν θα είχα ζητήσει το λόγο. Αλλά στον κανονισμό έχουμε το δικαίωμα να αντιδράσουμε όταν ε, αναφέρεται το όνομά μας. Δεν είναι νέος γύρος συζήτησης αυτό. Έτσι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για τους συναδέλφους. Ε, η κυρία Βεζιά ανέφερε το όνομά σας ε, πράγματι. Ευχαριστώ. Και συγγνώμη αν δεν σας έδωσα το λόγο. Έχετε δίκιο. Οπότε. Προθεσμοί για τροπολογίες ε, τώρα για αυτή την έκθεση 16 Ιανουαρίου 4 η ώρα. Ευχαριστώ λοιπόν τους ε, συναδέλφους. Πριν τις ψηφοφορίες λοιπόν, συναδελφοί, έχουμε άλλο ένα θέμα. Οι ψηφοφορίες είναι στις 11. Το τελευταίο θέμα είναι το σημεία 11 και 12 ε, Συγητής είναι ο κ. Ιγκουάνο και αφορά την σύναψη συμφωνιών ε, με την Βραζιλία. Δύο προτάσεις. Ο κ. του ΕΛΚ είναι συγητής και για τα δύο. Κύριε Σουγκουρεάνου. Ευχαριστώ. Δύο σχέδια συστάσεων για προτάσεις ε, συμφωνιών του Συμβουλίου, αποφάσεων του Συμβουλίου που τροποποιούν τις συμφωνίες μας με, τις, ε, με την ε, Βραζιλία για αυτούς που έχουν κανονικά διαβατήρια και αυτούς που έχουν διπλωματικά, υπηρεσιακά ή επίσημα διαβατήρια. Από τον Οκτώβριο του 2013. Η μέγιστη διάρκεια της παραμονής είναι 90 μέρες καθιαδήποτε περίοδο 180 μέρες. Τώρα γινόμαστε πολύ πιο συγκεκριμένοι. Η διάρκεια είναι μέρες και όχι μήνες. Και ο όρος από την ημερομηνία πρώτης εσόδου που δημιουργούσε πολλές ε, αμφιβολίες καταργήθηκε για να εφαρμόσουμε τον νέο ορισμό του τι είναι σύντομη παραμονή, τον Ιούλιο του 2014 η Επιτροπή ενέκρινε μια σύσταση για μια αποφαστού Συμβουλίου για να εγκρίνεται, για να εγκριθεί η έναξη διαπραγματεύσεων για να τροποποιηθεί η κατάργηση θεωρήσεων για σύντομες ε, παραμονές και το Συμβούλιο μπορεί να εγκρίνει την απόφαση αυτή μόνο εάν ο μόνο εάν το Κοινοβούλιο ε, δώσει σύμφωνη γνώμη. Εγώ ως συγητής προτείνω να δώσουμε τη σύμφωνη γνώμη και για τις δύο αποφάσεις. Κάτι ακόμη. Δεν λάβαμε την επίσημη νομική αίτηση από το Συμβούλιο και χωρίς αυτήν δεν μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία. Οπότε πείτε μα, πότε θα μα στείλετε αυτή την ε, αίτηση, το αίτημα το οποίο το περιμένουμε τόσο καιρό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και ο πρόεδρο, κύριε Ουγγουρεάνου. Θέλει κανεί το λόγο. Όχι, κανεί. Προθεσμία για τροπολογίε 14 Ιανουαρίου. Ευχαριστώ κύριε Ουγγουρεάνου. Ευχαριστώ για τι επεξηγήσει σα. Ευχαριστώ λοιπόν. Λοιπόν, στις 11 θα ψηφίσουμε. Διάλειμμα μέχρι τότε. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε. Ευχαριστώ.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

Uh, Παρακαλώ καθίστε. Είναι ηλεκτρονικέ ψηφοφορίε. Παρακαλώ να έχετε και τι κάρτε σα, αν δεν τι έχετε, να πάτε στον τρίτο όροφο να την πάρετε. Για όσου αναπληρωματικού δεν έχουν τι κάρτε του εδώ. Τι ήθελε να τα ακούσει. Ναι. Λοιπόν, όσο κάθεστε. Να επαναλάβω ότι είπα νωρίτερα. Όταν συζητούσαμε τους τριμερείς διαλόγους, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συμμετέχουν ε, στον ε, αριθμό ρεκόρ ε, τριμερών διαλόγων που γίνονται τώρα με ευθύνη της Επιτροπής μας. Να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μας, τους συνεργάτες των πολιτικών ομάδων. Είναι τρομερή δουλειά που θα έχουμε τους επόμενους τρεις-τέσσερις μήνες. Σας ευχαριστώ όλους που εργάζεστε τόσο σκληρά. Λοιπόν, έχετε καθίσει όλοι. Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Βλέπω ότι οι ορισμένοι χασμουργιούνται, αλλά επέμπτη είναι. Εντάξει, λοιπόν, συνάδελφοι, πρώτη ψηφοφορία. Απαλλαγή για την εφαρμογή του προπολισμού της Ένωσης για τους οργανισμούς ε, για το οικονομικό του 17. Απόδοση, οικονομική διαχείριση και έλεγχος. Εισηγητής είναι ο κύριος Φραντς. Κύριε Φραντς, θέλετε να πάρετε το λόγο πριν ξεκινήσουν οι ψηφοφορίες. Όχι. Ωραία. Περνάμε στις προφορίες. Ωραία. Συμβαστική 1. Άρχεται. πέρασε Δεκτή. Συμβαστική 2. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 6. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική 3. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 10. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Έχετε καθίσει όλοι. Τελική ονομαστική. Άρχεται. Πέρα. Δεκτή. 43 τρεις, ε, ε, κατά και 3 αποχές. Συγχαίρουν τον εισηγητή. Και να περάσουμε τώρα στην επόμενη ψηφοφορία. Και πάλι ε, Φραντς, εφαρμογή του προπολογισμού της ε, Ένωσης για τον οργανισμό Europol. Συμβαστική 1. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 2. Άρχεται. Πέρας. Ναι, τροπολογία 2. Και ψήφισα αντίστροφα. Mm. Αλλά εγκρίνεται. Τι πρόβλημα υπάρχει? Ναι, ναι. Ναι, εγώ κάτι έκανα λάθος, αλλά... Αλλά κάνω πολλά λάθη. Είναι μόνο ένα αυτό. Συμβαστική 2. Έχω, έχω. Κάνω πολλά λάθη. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 6. Τροπολογία 6. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική 3. Άρχεται. Πέρα. Δεκτή. Και τελικά η 11. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Τελική ονομαστική άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται 43 ψήφοι υπέρ, 2 κατά και μία αποχή. Επόμενο θέμα. Και πάλι ο κύριος Φραντς για τη Eurojust. Τροπολογία 1 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική 1 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 5. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική 2. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Τελική ονομαστική άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται 43 ψήφοι 2 κατά μία αποχή. Και τώρα πάμε στο επόμενο θέμα. Και πάλι Φράντς. Frontex. Συμβαστική 1 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Σημαστική 2 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Σημαστική 3 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική 4. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 10. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 11. Άρχεται. Αυτό Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική 5. Άρχεται. Πέρας. Δέκτη. Τροπολογία 15. Άρχεται. Πέρα. Απορρίπτεται. Τροπολογία 16. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται και αυτή. Τελική ονομαστική άρχεται. Πέρας. Δεκτή 42 ψήφι πέρι, 2 κατά 3 αποχές. Επόμενο θέμα του κυρίου Φραντς, ε, Οργανισμός Θεμελιδών Δικαιωμάτων Τροπολογία 1 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική 1 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική 2 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 8 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 9. Ε, ναι, άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 10. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 11. Άρχεται. Πέρας. Επίσης δεκτή, τελική ονομαστική άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται τα δύο ψηφί, πέτρες κατά μία αποχή. Επόμενο θέμα. Το κέντρο για τα ναρκωτικά. Φραντς, τροπολογία 1, άρχεται. Πέρασε. Δεκτή. Τροπολογία 2. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 3. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Και τροπολογία 4. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή και τελική ονομαστική άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται το κείμενο 43 ψήφοι υπέρ, 2 κατά μία αποχή. Και το επόμενο, Φραντς Σίπολ. Τροπολογία 1, άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 2, άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική 1. Άρχεται. Γιατί... Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 6. Ε, άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 8. Ε, συγγνώμη, συμβαστική 2. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 11. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 12. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Τελική ονομαστική άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται 45 ψηφιπέρ, 2 κατά και 0 αποχές. Και τέλος. Εάσο. Και πάλι Φραντς. Τροπολογία 1. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 2. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 3. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 4. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 5. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 6. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 8. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή Απορρίπτεται, συγγνώμη. Συμβαστική 1 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Και τροπολογία 12 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Και η τελική ονομαστική άρχεται. Πέρας και εγκρίνεται σαν δύο ψήφοι υπέρ, δύο κατά και μία αποχή. Και τώρα η Γιουλίσα. Φραντς και πάλι. Τροπολογίες 1 και 2, ταυτόσιμες, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρασε. Δεκτές. 3. Άρχεται. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 5 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 1 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 8 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 2 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική 3 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Και η τροπολογία 18 άρχεται. Πέρας. Δεκτή και αυτή. Τελική ονομαστική. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται 44 ψηφί υπέρ, 3 κατά 0 αποχές. Πάμε τώρα στην, στον Ευρωπαίο υπόπτη για τα, την προστασία των δεδομένων του κ. Φραντ πάλι, τροπολογία 1, άρχεται. Α, την αποσύρατε. Να συνεχίσουμε. Δεν χρειάζεται αν δεν θέλετε. Σαν ε, τα βιβλία του Κάφκα. Ψηφίστε το απλώς. Ένα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ποιος ξέρει γιατί. Δύο υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τρία. Πέρας. Εγκρίνεται. 4 έρχεται Πέρας. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, ονομαστική. Πέρας. Εγκρίνεται. 43, 3, μία αποχή τελευταία απαλλαγή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εκτελεστικοί Οργανισμοί, τροπολογία 1. Κύριε Μπόνη, έγινε λάθος στην παράγραφο 4, όταν ψηφίσαμε στην παράγραφο 4. Έχω αρνητικό πρόσωπο από την ομάδα, αλλά εγώ έβαλα συν. Στείλτε το σου για να σημειωθεί. Άλλαξε το αποτέλεσμα της προφορίας όχι, αλλά άμα θέλετε στείλτε το και γραπτός. Θα το συμπεριλάβουμε στα πρακτικά. Θα μπει στα πρακτικά μόλις το λάβουμε. Απλώς δεν θα αλλάξει έτσι καλλιώς η έκβαση της ψηφοφορίας. Πάμε πάλι στην Επιτροπή και Εκτελεστικούς Οργανισμούς, τοπολογία 1. Αυτό δεν ψηφίζαμε. Άντε να το ξανακάνουμε. 1. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Οκτώ άρχια η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τελική ψηφοφορία ονομαστική. Πέρας. Εγκρίνεται 44, 3, καμία εποχή. Συγχαρητήρια κύριε Φράνς για όλη σας τη δουλειά, για όλους αυτούς τους φακέλους. Uh, Συνάδελφοι, πάμε στην επόμενη έκθεση. Υλοποίηση των διατάξεων της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Μαρτίνα Άντερσον. Θες το λόγο Μαρτίνα πριν την ψηφοφορία. Πάμε απευθεία στην ψηφοφορία. Τροπολογία 37. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτω. 38. έρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 36. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 40. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 50. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 57 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 51 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9. Πέρας. Εγκρίνεται. 55. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 58. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 61. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 68. Πω πω, με συγχωρείτε, συμβαστική 10. Συμβαστική 10, ξέχασα όλη τη συμβαστική. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 68 άρχεται πέρας εγκρίνεται συμβαστική 11 άρχεται πέρας εγκρίνεται 75 άρχεται πέρας εγκρίνεται με τηλεοκές αναφορές 1 Α, όλες μαζί Ωραία ιδέα 1 ως 7 έρχεται η ψηφοφορία 1 ως 7 Όχι κόλπα ε, Πέρας Αυτό είπατε Εγκρίνεται Αιτιολογική σκέψη. 1. Συμβαστική 1. Πέρα. Εγκρίνεται. 12. Άρχεται. Πέρα. Εγκρίνεται. 13. Άρχεται. Εγκρίνεται. 2. Συμβαστική 2. Πέρας. Αγκρίνεται. 19. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 21. Άρχεται. Όχι, αυτά δεν γίνονται όλα μαζί. 19. Πέρας. Εγκρίνεται. 23 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 25 υπέρ. Μάλλον έρχεται, ε, να για μισό λεπτό. Έχετε δίκιο, μπορούσαμε να τα είχαν κάνει unblock. Όχι, όχι, δεν μπορούσαμε, δεν μπορούσαμε. Πέρας, εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 5. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 29. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ονομαστική. Πέρας. Εγκρίθηκε με 40 ψήφου υπέρ, τα κατά και 0 αποχές. Συγχαρητήρια. Στον εισηγητή, στην εισηγήτρια Μαρτίνα. Α, εντάξει, καλά τα έκανα, ωραία. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια. Επόμενη ψηφοφορία. Μάμικινς εμπορία και χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών. Κύριε Μάμικιν, θέλετε να πείτε κάτι? Όχι, ψηφίζουμε. Ωραία, μία ψηφοφορία. Άρχεται. Α, όχι, μια στιγμή. Ε, έναρξη των διοργανικών διαπραγματεύσεων. Τι θέλει. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 45 ψήφι υπέρ, 2 κατά καμία αποχή. Συγχαρητήρια, Ανδρέη. Πρώτος διάλογος στις 21 Ιανουαρίου. Και τώρα περνάμε στην εφαρμογή των διατάξεων συνθήκης για την ενισχυμένη συνεργασία έκθεσης Δεχόφσκι. Μπορούμε να περάσουμε στη ψηφοφορία. Τόμας, θέλεις τον λόγο? Θέλεις. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω όλους. Καλή χρονιά. Μπορούμε να ψηφίσουμε. Ωραία. Καινοτόμο αυτό. Ευχαριστούμε. Ωραία, είχα την ευκαιρία να βρω και τον κατάλογο των ψηφοφοριών. Τροπολογία 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Δεκτή. 14 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 15 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 16 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 18 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 21. Α, όχι 19. 19 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 20 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Η 21 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 22 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. απορρίπτεται η 27 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται η 28 άρχεται η ψηφοφορία όχι 28 και είναι δικιά σας κιόλας μόνικα. ψήφισαν όλοι πέρας απορρίπτεται ε, συγγνώμη η 29 άρχεται ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται συμβαστική 2 άρχεται ψηφοφορία πέρας δεκτή 32 άρχεται ψηφοφορία πέρας δεκτή εκτιμώντας ε, τροπολογία 1 αρχή ψηφοφορία πέρασε απορρίπτεται συμβαστική 3 αρχή ψηφοφορία πέρασε δεκτή τροπολογία 2 αρχή ψηφοφορία πέρασε και απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 9. Ε, ναι, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Επίσης απορρίπτεται τελική ψηφοφορία ονομαστική. Άρχεται. Και πέρας. Και δεκτή. 36, 6 κατά, 3 εποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία. Εφαρμογή της Χάρτας των Δικαιωμάτων στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης. Ο κύριος Ντεγιόγκ είναι ο εισηγητής. Θέλετε τον λόγο? Όχι. Περνάμε στην ψηφοφορία. Τροπολογία 19. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. απορρίπτεται 20 και 21 ταυτόσημες άρχεται ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 22 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 23 άρχεται ψηφοφορία πέρας Επίσης απορρίπτεται. Ε, συμβαστική 2 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική 1 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 29 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. δεκτή 33 αρχιτή ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 34 αρχιτή ψηφοφορία πέρας δεκτή 35 αρχιτή ψηφοφορία Πέρας. Απορρίπτεται. 36 άρχεται Πέρας. ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται 37 άρχεται η ψηφοφορία. Δεκτή. 30, όχι. συγγνώμη, συμβαστική 3. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 44. Δεκτή 45 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε δεκτή 46 αρχιτή η ψηφοφορία πέρας δεκτή 48 αρχιτή η ψηφοφορία πέρας δεκτή 49 αρχιτή η ψηφοφορία πέρας δεκτή 50 αρχιτή ψηφοφορία. Πέρασε. Δεκτή. 51 αρχιτή ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 52 αρχιτή ψηφοφορία. Πέρασε. Δεκτή. 53 αρχιτή ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 54 αρχιτή ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή 55 αρχιτή ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή 57 αρχιτή ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή 63 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 64 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. δεκτεί 65 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 66 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 67 άρχεται η ψηφοφορία πέρας δεκτή. Αιτιολογικές αναφορές. Ένα με 4 μπορούμε να τις κάνουμε μαζί. Όχι. Ναι. Τροπολογία 1. Αρχιετή ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 2. Αρχιετή ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 3, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 4, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Εκτιμώντας, τροπολογία 5, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 6, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 7 άρχιδη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 8 και 9 ταυτόσιμες άρχιδη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Ταπολογία 10 άρχιδη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 11 και 12 ταυτόσημες. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 13 και 14 ταυτόσημες. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Επίσης απορρίπτεται 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. τι ναι, 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. απορρίπτεται 18 τι είναι 18 Αρχιετή ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται και τελική ονομαστική ψηφοφορία Αρχιετή ψηφοφορία πέρας δεκτή 39 ψήφους 8 κατά καμία αποχή Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Στον ευχαριστώ. Uh, και το επόμενο θέμα. Έκθεση Μακοβέη. Οι έρευνες που κάνει η Όλαφ όσον αφορά τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την αποτελεσματικότητα των ερευνών της Όλαφ. Κυρία Μακοβέη, θέλετε να πάρετε το λόγο πριν την ψηφοφορία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους και τους κοιόδες να διευκρινίσουμε τη σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και της Όλαφ είναι σημαντικό για να μην υπάρχει επικάλυψη και να λειτουργεί καλά η ανταλλαγή πληροφοριών για να λειτουργήσει καλύτερα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Α, τροποποιούμε τους κανόνες δηλαδή της Όλαφ για να τους προσαρμόσουμε στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, λέει Ψηφίζουμε. Τροπολογία 51. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 52. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Ε, συμβαστική 5. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 59 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 63 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 64 άρχεται. Πέρασε. Δεκτή. 65 άρχεται. Πέρασε. Απορρίπτεται. 66 άρχεται. Πέρασε Δεκτή. 67 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 68 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 7 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 69 άρχεται. Πέρας. δεκτή 70 άρχεται πέρας δεκτή συμβαστική έξι, άρχεται πέρας δεκτή 72 άρχεται πέρας δεκτή 73 άρχεται πέρας δεκτή 76 άρχεται πέρας δεκτή 77 άρχεται πέρας δεκτή 78 άρχεται πέρας δεκτή συμβαστική 6α άρχεται πέρας δεκτή 82 άρχεται πέρας Δεκτή. 81 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 83 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 84 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 85 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 86 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 87 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική 7 άρχεται. Πέρας. δεκτή. Συμβαστική 8 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 91 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 94 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική 8α άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 11 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 97. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 98. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική ενέργεια Πέρας. Δεκτή. Δεκατέσσερα. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Εκατόν δύο. Άρχεται. Πέρασε. δεκτή. Δεκαπέντε άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Σημαστική δέκα άρχεται. Πέρας. Δεκτή 17 άρχεται. Πέρας. Δεκτή 107 άρχεται. Πέρας. Δεκτή 108 άρχεται. Πέρας. δεκτή συμβαστική 11 άρχεται πέρας δεκτή 113 άρχεται πέρας δεκτή 114 άρχεται πέρας δεκτή 115 άρχεται Πέρας. Δεκτή. 116. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Αιτιολογικέ σκέψει. Τροπολογία 20. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 21. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 22. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 23. Άρχεται. Πέρας. Πέρας δεκτή. 24. Άρχεται. Πέρα. Α, πέρασε. Δεκτή. 25 άρχεται. Πέρασε. Δεκτή. Συμβαστική 1 άρχεται. Πέρασε. Δέκτη. Συμβαστική 2 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 35 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική 3 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική 4 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Τραπολογία 40. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 41. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 42. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 43. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 44. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 45. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 46. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 47. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 48. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 49. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 50. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τελική ονομαστική. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 40 ψήφοι υπέρ, 4 και μία απογεία συγχαίρουμε τον εισηγητή. Και μία τελευταία. Μία ενιαία ψηφοφορία η καταπολέμηση της απάτης και της παραχάραξης ε, ε, μεθόδων πληρωμών χωρίς νομίσματα ή χαρτονομίσματα. Η Σιλβί Βον Κάουφμαν δεν είναι παρούσα. Ψηφίζουμε λοιπόν η σιλβι βον καουφμαν δεν παρουσα ψηφοφορία για ε, τις διοργανικές διαπραγματεύσεις. Μία νέα ονομαστική η οποία και άρχεται. Πέρας. 45 πέρα, μία ψήφος κατά και καθόλου απογεύση. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ για την υπομονή σας. Ε, ήταν ε, πολύ μακριά η ψηφορία. Και είναι και το τέλος της συνεδρίασής μας. Δεν υπάρχουν άλλα θέματα. Θα τα ξαναπούμε στις 23 Ιανουαρίου. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.